Good afternoon, everybody. Um, we'll recommence the, the meeting. I, I was waiting a few moments, hoping that a few more of the shadows... Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε, αλλά θέλαμε να έχουμε και τους σκιώδεις εδώ πριν ξεκινήσει η συγγήτρια. Είμαστε στο σημείο 16 τώρα της ημερήσιας διάταξης το θέμα τη ε, Ελίζα Φεραίρ είναι έκθεση Πρωτοβουλία για τη διαχείριση της διασυνοριακή κρίσης στον τραπεζικό τομέα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, τώρα θα δούμε τις τροπολογίες. Ελίζα, έχεις το λόγο. Thank you very much, Sharon. Um, Eh, eh, η έκθεση δέχτηκε 247 τροπολογίες, συν 12 από την ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η γενική μου εκτίμηση για αυτές ε, τις ε, τροπολογίες είναι πως εν γέννη είναι πολύ θετικές και προσδίδουν αξία στο κείμενο. Προσθέτουν. Αυτό είναι το γενικό μου σχόλιο. Τώρα, για να μπω σε πιο συγκεκριμένε λεπτομέρειε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ποια είναι η φιλοσοφία που διέπει την πρόταση. Η φιλοσοφία αυτή είναι ότι το Κοινοβούλιο πρέπει μέσω αυτής της πρότασης να διαβιβάσει μια έννοια, μια ιδέα πολύ, πιο, πολύ στεναρή και ξεκάθαρη ότι δηλαδή μετά από την κρίση και μετά από τα όσα συνέβησαν στις ε, οικονομικές αγορές τελικά καταφέραμε να διατηρήσουμε την εσωτερική μας αγορά όμως ε, και μπορέσαμε όλα τα κράτη-μέλη να μοιραστούν τα πλεονεκτήματα αυτής της εσωτερικής αγοράς ε, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το moral hazard, ότι η διαχείριση της κρίσης ε, δεν μπορεί να είναι ένα bailout, ή ένας τρόπος ε, για να έχουμε μία ασφάλεια σε περίπτωση λιγότερο προσεκτικής διαχείρισης και άρα θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρος ο βασικός στόχος τον οποίο προτείνουμε. Στόχος είναι να διευκολύνουμε να την, ε, το κλείσιμο ή τη χρεοκοπία μιας τράπεζας ή την απομόνωση μιας τράπεζας πριν αυτή να μεταδώσει την, ε, το πρόβλημά της και σε ολόκληρο τον τομέα. Αυτό που μπορούμε δηλαδή να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα ταμείο, να αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση και σταδιακά να εργαστούμε στην κατεύθυνση της σύγκλησης της νομοθεσίας. Αλλά αντιλαμβανόμενοι ότι δεν μπορούμε να πνίξουμε τις αρχές και κυρίως την τραπεζική αρχή που έχει δημιουργηθεί με, μια, ε, με πολυάριθμα προβλήματα. Διότι εμείς ε, συμφωνούμε με τις τράπεζες και με το θεσμικό όργανο ότι αποτελούν έναν μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο και που άρα θα πρέπει πριν από όλες τις άλλες να είναι συντονισμένες ε, και να επιβλέπονται με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές αρχές που προτείνουμε. είναι αυτές αρχές οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συνδυάστηκαν ή διατυπώθηκαν και στο πλαίσιο της έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή που συνέταξε ο συνάδελφος Γκαρσία Μαρσάλη. Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο σημείο. Σε αυτή τη φάση είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση και το μήνυμα του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρό και φιλόδοξο διότι θα μπούμε σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων όπου δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα να προχωρήσουν ε, χωρίς να έχουμε συγκεκριμένο στόχο και φιλοδοξία. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο όλα αυτά να τα διαβεβαιώσει, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση απέναντι στις εντάσεις και στις ε, άκαμπτες θέσεις του Συμβουλίου. Και νομίζω πως θα εξυπηρετήσουμε την Ευρώπη αν είμαστε συνεπείς και φιλόδοξοι. Μεγάλο κομμάτι των τροπολογιών που υποβλήθηκαν νομίζω πως χάνουν το νόημά τους εάν λάβουμε υπόψη την διακοινοβουλευτική συμφωνία που ήδη καταφέραμε να έχουμε για την ψήφιση της έκθεσης Γκαρσία Μαργκάλιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή γνώμη μου είναι ότι το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει πολύ συνεπή θέση και να συγκλίνουν οι διάφορες εκθέσεις με συντονισμένο τρόπο ώστε να μην είναι η θέση μας ε, κατακαιρματισμένη ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές ομάδες και τους τις διάφορες εκθέσεις. Στην περίπτωση της έκθεσης ε, του Γκαρσία Μαργκάλιο, κάναμε προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις και δεχτήκαμε τις εξής αρχές. Πρώτον, αρχές. Πρώτον, ορίσαμε ποιες είναι οι τράπεζες που έχουν συστημικό χαρακτήρα. Και η ορολογία, και θα τα πω στα αγγλικά για να μην έχουμε ε, μπερδέματα, δέχτηκε αυτή την ιδέα για τις τράπεζες, δηλαδή που θα μπουν σε αυτό το ειδικό καθεστώς, Cross-border systemic banks είπαμε, δηλαδή οι τράπεζες πρέπει να είναι cross-border και πρέπει να είναι και συστημικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν μία διάσταση ή μία περιπλοκότητα ή μία διασύνδεση που τις μετατρέπουν σε τράπεζες πιο περίπλοκες, περίπλοκου χαρακτήρα από ό,τι άλλες και άρα και πιο επικίνδυνο να εισάγουν ε, προβλήματα στο σύστημα και άρα τράπεζες που χρειάζεται να τις παρακολουθούμε μεγαλύτερη προσοχή και κατά προτεραιότητα. Δηλαδή είναι οι τράπεζες αυτές που αποκαλούμε fast track. Η δεύτερη αρχή ήταν να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή η ευθύνη η ευθύνη η μεγαλύτερη για την εποπτεία όχι, ε, που είναι αυτόνομη λειτουργεί ως ένα συλλογικό όργανο σε συνεργασία με τα cross border stability groups αλλά είναι υπεύθυνο για διαχείριση κρίσης σε περίπτωση ε, ε ξεσπάσει και σε συνεργασία με τους ε, ηγέτες, τους διευθυντές μάλλον των cross border systemic banks. Επίσης, ε, αποφασίσαμε για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Σταθερότητας. Είναι ένα ξεχωριστό ε, ταμείο με το Deposit Guarantee Scheme για την εγγύηση δηλαδή των καταθέσεων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί καταρχήν σε μια πρώτη φάση από τις συστημικές τράπεζες με βάση την εκτίμηση του κινδύνου που αυτές εισάγουν στο σύστημα. Δηλαδή, αν μια συστημική τράπεζα έχει ε, λειτουργίες χαμηλού κινδύνου, θα πρέπει να συμβάλλει κατά πολύ λιγότερο σε αυτό το ταμείο από ότι μια άλλη τράπεζα που έχει λειτουργίες και ε, συναλλαγές υψηλού κινδύνου. Τέταρτο, αυτό που συμφωνήσαμε ήταν να έχουμε μια, ένα ψήφισμα, ε, να δημιουργήσουμε μια, ένα task force μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, ώστε να μπορεί να παρέμβει κατεπηγόντως σε περίπτωση που μια τράπεζα αντιμετωπίζει προβλήματα. Αυτές οι τέσσερις γραμμές λοιπόν ε, χαρακτήριζαν όλες μας τις εργασίες ε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και την προπαρασκευή για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και επίσης προς αυτή την κατεύθυνση εργαστήκαμε με τους σκιώδεις εισηγητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων και για την προπαρασκευή αυτής εδώ της συνεδρίασης και υπήρξε σύγκληση ανάμεσα σε όλους ότι όντω η θέση του, του Κοινοβουλίου ήταν πιο συνεπής και σταθερή αν όντω ε, εμεί υιοθετούσαμε αυτού του είδου τι αρχέ. Αν όντω γίνει αυτό, πολλέ από τι τροπολογίε που έχουν υποβληθεί προ την δική μου έκθεση καταπίπτουν διότι δεν έχουν πλέον νόημα. Όπως κατέπεσαν εξάλλου και στην περίπτωση της έκθεσης του Γκαρσία Μαργκάλιο. Και αν υπάρχει αυτή η συνοχή, γύρω στις 200 από τι 47 καλύπτονται από αυτήν την γενική συμβιβαστική συμφωνία. Αν όντως συμβεί έτσι, οι υπόλοιπε τροπολογίε είναι τροπολογίε τι οποίε εγώ θα τοποθετούσα στι εξή διαστάσει. Υπάρχει δηλαδή μία συγκεκριμένη τυπολογία. Ο πρώτο είδο ε, τροπολογιών είναι αυτέ οι οποίε εμπίπτουν σε μία εθνική λογική και γι' αυτό νομίζω ότι δεν εμπίπτουν εδώ σε αυτήν εδώ την έκθεση. Δηλαδή δεν καλύπτονται από τη Γενική Συμβιβαστική Συμφωνία αλλά δεν εμπίπτουν μέσα στην ε, έκθεση γιατί είναι εκτό του πνεύματο αυτού που θέλουμε να πετύχουμε στο Κοινοβούλιο. Είναι, υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες ε, προτείνουν ε, τεχνικές ε, και νοηματικέ βελτιώσει. Αυτές είναι ενδιαφέρουσε περισσότερες και θέλω μόνο να κάνω μια παρατήρηση για μια σειρά από τι προτάσει που έχουν υποβληθεί κυρίως από την συνάδελφο Σουίνμπεργκ όπου προσπαθεί να ευθυγραμμίσει την θέση της Ευρώπης με τη διεθνή θέση. Εγώ νομίζω ότι αυτές είναι σκέψεις τις οποίες μπορούμε να απορροφήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ελπίζουμε πως οι διεθνείς πρωτοβουλίες θα φτάσουν σε τόσο πολλές λεπτομέρειες ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν πως υπάρχει δυνατότητα να γίνουν κάποιες προτάσεις σύγκλησης, αλλά χωρίς να αποκλείουμε ή μάλλον χωρίς να υποχρεώνουμε την απόλυτη ταύτιση. Δηλαδή το διεθνές πλαίσιο να σταθεροποιηθεί για να κάνει μετά η Ευρώπη κάτι. Η Ευρώπη πρέπει να είναι διεθνής εταίρο και να προσπαθήσει να βοηθήσει στο σχηματισμό του διεθνούς πλαισίου. Ένα άλλο είδος τροπολογιών είναι αυτές οι οποίες ε, μπαίνουν σε υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά την πρόταση μέτρων ή συγκεκριμένες προτάσεις ε, για το ποια θα είναι τα μέτρα ε, τα μέσα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Πιστεύω πως αυτά τα μέτρα, σε αυτό το βαθμό λεπτομέρειας δεν, εγώ δεν έχω αντίρρηση επί της αρχής, αλλά νομίζω πως αποσταθεροποιούν την έκθεση, διότι είναι μια έκθεση πολιτικού μηνύματος και, να σε, και θα πρέπει να υπάρχει το ίδιο επίπεδο λεπτομέρειας σε ολόκληρη την έκθεση. Γι' αυτό και το να μπούμε σε εξαιρετικά πολλές λεπτομέρειες σε κάποια μονοσημεία, αναιρεί το νόημα του μηνύματος που θέλουμε εμείς να διαβιβάσουμε. Γι' αυτό εδώ θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες συμβιβαστικέ τροπολογίες. Υπάρχουν και άλλες κάποιες τροπολογιών που είναι διευκρινιστικές και πάλι, πιο λεπτομερείς. Ε, ε, επί της αρχής νομίζω πως πρέπει να ενσωματωθούν Ο Όλη Σμιτ και ο Σβέν Γκίγκολτ έκαναν κάποιες τέτοιες προτάσεις που βελτιώνουν το κείμενο. Από πλευρά των άλλων συναδέλφων και από την Ταρνούτα Χούμπνερ έχω κάποιες τέτοιες τροπολογίες. Αν λοιπόν ξεκαθαρίσουμε και σκεφτούμε όλα αυτά τα είδη των τροπολογιών και εδώ ολοκληρώνω, προσπαθώ και Ήδη έχω κάποιες συμβαστικέ προτάσεις που προσπαθούν να είναι όσο γίνεται πιο διευρυμένες και να καλύψουν το μεγαλύτερο τμήμα των τροπολογιών που έγιναν γιατί εκεί όπου υπάρχει δυνατότητα να υπάρξουν συμβιβαστικέ τροπολογίε θα το κάνω και να έχουμε ένα, μια πολύ περιορισμένη, ένα πολύ περιορισμένο σύνολο τροπολογιών, 10-12, για αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα. Ή είναι αντίθετες στο πνεύμα ή είναι νόμιμες και θεμητές ή εναλλακτικά μπαίνουν σε τόσο πολλές λεπτομέρειε που πιστεύω πως δεν θα επιτρέψουν συνένεση, αλλά και δεν βοηθούν, δεν προσθέτουν τίποτα στα μηνύματα και στις κεντρικές ιδέες. Γνωρίζουμε ότι σε αυτή τη φάση οι διαπραγματεύσεις τόσο στο επίπεδο του τριμερούς διαλόγου, τον οποίο δεξάγει ο συνάδελφος Γκαρσία ε, ε, Μαργάλιο, όσο και νέα πρωτοβουλία από πλευρά τη Κομισιόν ε, βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά πιστεύω πως από πολιτική άποψη θα πρέπει να έχουμε μια συμπαγή και σταθερή θέση ως Κοινοβούλιο και να μπούμε στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο μιας γενικής κοινή γραμμής. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρότεινα να συντάξω συμβιβαστικέ τροπολογίε, τι οποίε αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέλιξη, υπό προετοιμασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Κάρα, εσεί θα μιλήσετε ε, αντί τη κυρία Τούμπνερ. Ε, πραγματικά αντικαθιστώ την Τανούτα Χούμπνερ, την σκιώδη συγγήτριά μας είμαι σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚ και εγώ έχω κάποιες αμφιβολίες για τη διάκριση μεταξύ συστημικών και μη συστημικών τραπεζών. Έχω ορισμένε αμφιβολίες επ' αυτού. Αυτό ήδη ήταν ένα μεγάλο θέμα όταν αρχίσαμε την εργασία μας πάνω σε αυτήν την έκθεση. Μία διάκριση μεταξύ συστημικών και μη συστημικών θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λύσει. Αν χρησιμοποιήσουμε ποσοτικά κριτήρια, τότε ε, η διαδικασία ορισμού της φύσης των τραπεζών ε, θα είναι λυπής, δεν θα είναι σωστή. Διότι θα πρέπει να καθορίσουμε ποσοτικά πότε η τράπεζα σταματά να είναι συστημική ή πότε ξεκινά να είναι συστημική. Εάν κολλήσουμε ετικέτες σε τράπεζες και τις ονομάσουμε συστημικές, θα νομίσουν ότι είναι τόσο πολύ σημαντικές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ώστε να έχουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι ό,τι και να κάνουν οι αρμόδιες αρχές θα τις σώσουν. Δηλαδή θα πιστέψουν οι λεγόμενες συστημικές τράπεζες ότι είναι υπεράνω των άλλων τραπεζών. Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να αποκλίνουμε και να μην εφαρμοστεί ε, ακριβώς η αρχή του moral hazard πρέπει να υποστηρίξουμε τις τράπεζες οι οποίες ε, δραστηριοποιούνται είτε μέσω θηγατρικών είτε μέσω άλλων συνεργασιών. Ε, γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν οι επιφυλάξεις ε, όσον αφορά την ετικέτα του συστημικού. Η Ντανούτα Χούμπνερ επίσης πιστεύει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο σε βάθος τις διασυνοριακές συναλλαγές. Όσον αφορά δε την τροπολογία 124, αυτή η τροπολογία έχει ως στόχο την ελάχιστη παρέμβαση, την αντικατάσταση των μυστικών αρχών όσον αφορά την ε, διετερική μεταφορά κεφαλαίων, το Intra Group assets ε, transfers. Αυτές οι ενδοετερικές μεταφορές ε, πολλές φορές στοχεύουν στην αύξηση της ε, ρευστότητας της μητρικής εταιρείας, της έδρας, ε, στην έδρα της τράπεζας. Δεν θα πρέπει λοιπόν αυτές οι διετερικές, ενδοετερικές μεταφορές ενεργητικού να διακινδυνεύσουν τα κεφάλαια, τα επενδυμένα των καταθετών. Πρέπει να εξετάσουμε τις επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τη θέση των καταθετών ε, μέσω των εγγυήσεων καταθέσεων. Πιστεύουμε ότι αυτή η τροπολογία θα ανοίξει το δρόμο για μια ισόρροπη κατανομή του βάρους, της ευθύνης και της κατανομής του κόστους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου, διότι όλη η διεθνής πτυχή δεν λαμβάνεται υπόψη στο κείμενο. Πιστεύω ότι ορισμένα από τα σχόλια των G20 να γίνουν αποδεκτά και να ενσωματωθούν. Ιδίω επειδή έχω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στην αξιολόγηση της διαφοράς μεταξύ μιας διασυνοριακής τράπεζας και των άλλων. Μερικές διασυνοριακές ε, τράπεζας δεν είναι ενδοκινοτικά διασυνοριακές, αλλά διασυνοριακές ως προς άλλες χώρες, ως προς τρίτη επικράτεια. Ίσως λοιπόν εμείς εδώ εξετάζουμε την ουρά του σκύλου μόνο και όχι ολόκληρο το σκύλο. Γι' αυτό, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια σωστή διασυνοριακή διαχείριση, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι ορισμένοι μεγάλοι παίκτε μπορεί μεν να έχουν τεράστιες διασυνορικές συναλλαγές, αλλά δεν εδρεύουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ε, να καλύψουμε όλες αυτές, ε, όλα αυτά τα ιδρύματα, ιδίως μεγάλες τράπεζες που έχουν ε, μεγάλες συναλλαγές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω θηγατρικών αλλά και αλλού, στην Ασία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι λοιπόν όλες με ε, έχουν την έδρα του στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, διότι εδώ υπάρχει μία διεθνής ε, πτυχή. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Deutsche Bank, μην ξεχνάτε, ότι έχει περισσότερο αριθμό εργαζομένων στις ε, θηγατρικές παγκοσμίω από ό,τι στην έδρα της. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε ακριβώς ποιο ποσοστό του μεγέθους των συναλλαγών της τράπεζας γίνεται ε, ενδοκινοτικά και πιο έξω, ε, όχι ενδοκινοτικά. Η, βεβαίως εδώ περισσότερο μιλάμε για τις ε, διασυνοριακές ε, συναλλαγές των ε, τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεδομένου ότι ε, βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον πρέπει να δούμε πώς γίνεται η διαχείριση των, ε, του ενεργητικού και εξοκοινωτικά. Τώρα, για την ετικέτα της συστημικής ή μη συστημικής τράπεζας, ας μην ξεχνάμε ότι μία μεγάλη προβληματική τράπεζα δεν ήταν ούτε καν ε, είχε διασυνοριακές συναλλαγές, όμως αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση ως συστημική τράπεζα. Πώς θα ορίσουμε λοιπόν μία συστημική και όχι συστημική. Πρέπει να εξετάσουμε διαφορετικά κριτήρια και πιστεύω ότι αυτά που προτείνει η κυρία Χούμπνερ είναι σωστά. Είναι, είναι σωστά και τα υποστηρίζω. Ε, όσον αφορά τώρα την εκροή κεφαλαίων, ε, υπάρχει τεράστια εκροή κεφαλαίων ε, και υπήρξε και από τις θηγατρικές προς την Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης. Δηλαδή διαρροή κεφαλαίων διεθνώς, όπου κεφάλαια του ενεργητικού φύγαν, διέφυγαν από τις θηγατρικές. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε και εδώ τα ίδια κριτήρια απαγόρευσης και να πούμε ότι αυτές οι θηγατρικές, ή τράπεζες δεν θα επιτρέπεται να μετακινούν ε, τα, το ενεργητικό τους ε, αν δεν σέβονται συγκεκριμένους κανόνες. Υπάρχει λοιπόν η διεθνή πτυχή που εμπλέκεται εδώ. Εάν δεν αξιολογήσουμε πόσες από τις τράπεζες αυτές είναι πανευρωπαϊκές δασιενεργειακές. δεν θα κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση. Δεν μας αρκούν μόνο τα ε, ε, ευρωπαϊκά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε και διεθνώς πώς κινούνται αυτές οι τράπεζες. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και χρειάζεται και πάρα πολύ δουλειά και ευχαριστώ την εισηγήτρια, ε, ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια διότι ανέλαβε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο θέμα και έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ε, για να επιτύχει μια ευρεία συνένεση. Μπορεί να επιτύχει στο τέλος. Πού, ξέρουμε, μπορεί να αλλάξουμε τη γνώμη μας τελευταία στιγμή. Ελπίζω όμως όχι. Ε, ό, όταν θέλουμε να ορίσουμε τράπεζες που ενέχουν έναν συστημικό κίνδυνο ή διασυνοριακό κίνδυνο είναι σχεδόν αδύνατον. Αφήστε το λοιπόν. Πολλοί λένε αφήστε το, είναι αδύνατον. Μην το πιάνετε αυτό στα χέρια σας καθόλου. Δεν είναι όμως ε, αυτός ο σωστός τρόπος. Ε, πρέπει να κάτι να κάνουμε. Τουλάχιστον να βρούμε ορισμένες απαντήσεις σε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα. Εάν ε, η πρότασή μου είναι να περιοριστούμε στις ε, τράπεζες που έχουν διασυνοριακές συναλλαγές. Κάποιος μου λέει μπορεί να είναι 700 αυτές οι τράπεζες. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι 700, εγώ πιστεύω ότι είναι 44, 50, εκεί γύρω. Πιστεύω ότι δεν θα είναι σωστό να ε, έχουμε έναν ορισμό που να μας επιτρέπει να πούμε αυτό είναι συστημικό, αυτός ο κίνδυνος είναι συστημικός, εξού και η τράπεζα είναι συστημική. Εμείς μιλάμε για, για διασυνοριακές συναλλαγές, διασυνοριακές τράπεζες και αυτό προτείνει και η συγγήτρια προς το παρόν και μπορούμε να το δεχτούμε. Όχι ότι εδώ βρισκόμαστε στο τέλος ε, της πορείας μας, αλλά θα χρειαστούν και πολλά άλλα. Προς το παρόν όμως αρκεί αυτός ο ορισμός. Εν συνεχεία έχουμε αυτό το ταμείο. Το Ταμείο Δημοσιο... Ε, Δημοσιονομικής Σταθερότητας, ε, ε, Οικονομικής Σταθερότητας. But, uh, properly... Σταθερότητας. η διαχείριση του ταμείου αυτή μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμη. Ε, η Κομισιόν παίζει έναν ενδιάμεσο ρόλο. Πιστεύω ότι αυτή η πρόταση όμως για το ταμείο αυτό ε, είναι σωστή, Financial Stability Fund. Είναι ευρωπαϊκό ταμείο και μπορούμε να το δεχτούμε. Το ψήφισμα, άλλο ένα δύσκολο θέμα προτείνω το ψήφισμα να είναι ανεξάρτητο και να μην είναι συνδεδομένο στο ε, European Banking Agreement, στο EBA, e EBA. Διότι διαφορετικά, στο European Banking Authority, διότι διαφορετικά μπορεί να υπάρχει μια διασύνδεση που δεν είναι σωστή. Το ψήφισμα αυτό να μην συνδέεται λοιπόν με το EBA. Όσον αφορά τώρα τα μέσα, τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, Έχω την εντύπωση ότι η κυρία Φερέιρα πιστεύει ότι ορισμένες προτάσεις, ορισμένες τροπολογίες είναι υπερβολικά λεπτομερείς. Πιστεύω όμως ότι αυτό το μέσον πρέπει να προτείνει μια εναλλακτική λύση. Ε, πρέπει να δεχτούμε ορισμένα εναλλακτικά εργαλεία. μέσω τροποποίησεων. Γι' αυτό τι ζητώ ε, σε αυτό το toolbox, ε, σε αυτό το βαλιτσάκι με τα εργαλεία, το κουτί με τα εργαλεία, να δεχτεί ορισμένα συστατικά. Αναφέρθηκε επίσης και το θέμα των intra-group assets, δηλαδή των ε, ενδοετερικών, του ενδοετερικού ενεργητικού, των ενδοετερικών κεφαλαίων. Εδώ πιστεύω ότι αρκετοί από εμά συμφωνούν. Γενικά, κυρία εισηγήτρια, έχετε κάνει θαυμάσια δουλειά. Πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε μέχρι ενός βαθμού συνένεση. Είναι ένα λίγαν περίπλοκο θέμα. Ορισμένοι από εμά βεβαίω έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας σε αυτά που συμβαίνουν στις χώρες μας. Έχουμε πλέον εμπειρία και πιστεύω ότι από την εμπειρία τη δική μας, από τις χώρες μας, μπορεί να βγει κάτι καλό κάτι σωστό. Τα πασίματα μαθήματα λοιπόν. Πολλοί από εμά έχουν μάθει ότι για να προλάβεις μια κρίση πρέπει αυτό το, το βαλιτσάκι, το toolbox να έχει πάρα πολλά εργαλεία, πάρα πολλά μέσα τα, οποία μπορούν να εφαρμοστούν προληπτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ από τους σκιώδης. Πανέβασα από το κρατήριο χωρίς μικρόφωνο. Α, είσαστε Σκιώδης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η έκθεση αυτή για να αποφεύγονται οι πτωχεύσεις των μεγάλων τραπεζών και πρέπει να υπάρξει μια καλή πλαισίωση για την οικονομία, για τους πολίτες και τους φορολογούμενους. Έτσι λοιπόν ευχαριστώ και χαιρετίζω την κυρία Φερέρα για τη δουλειά της που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σημείο κίνησης και περιλαμβάνει και σημαντικά στοιχεία πρόοδου. Οι προτάσεις που κάναμε από πλευρά των Πρασίνων πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση και όντως έχουν σαν στόχο την πρόοδο σε δύο κυρίως πυλώνες. Πρώτα απ' όλα το Ευρωπαϊκό Ταμείο, τα Εθνικά Ταμεία συντονισμένα, έτσι όπως τα προβλέπουμε σήμερα, δεν πρέπει να θεωρούνται μια εγγύηση για τις τράπεζες από οποιοδήποτε κίνδυνο αντιμετωπίζουν για να αποφύγουν τη χροκοπία. Στη συνέχεια, μια τέτοια εγγύηση, ακόμα και αν χρηματοδοτείται από τις ίδιες τις τράπεζες, δίνει στις τράπεζες την εντύπωση ότι μπορούν να πάρουν όποιο κίνδυνο και να είναι, μια που έτσι κι θα καλύπτονται απριόρι. Αντί λοιπόν να ενισχύσουμε τη ρύθμιση των οικονομικών αγορών, αντίθετα την αποδυναμώνουμε. Η δεύτερη αρχή απορρέει από την προηγούμενη. Η έκθεση αυτή νομοθετικής πρωτοβουλίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο έπακρον. Πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να υιοθετήσουν νέα μέτρα όσο γίνεται πιο τολμηρά. Και πρέπει και εμείς, συνεπώς, να δείξουμε ότι είμαστε τολμηροί. Πρέπει οι κανόνες παρέμβασης των υποπτικών αρχών να καθορίζονται εξάντε, να είναι δεσμευτικοί. Αυτό σημαίνει κανόνες σχετικά με το όριο παρέμβασης, όπως επίσης και τους κανόνες που έχουν να κάνουν με την κατανομή του βάρους. Πώς γίνεται σωστά αυτή η κατανομή του βάρους όταν έχουμε να κάνουμε για διασυνοριακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, συστημική τράπεζα, πρέπει να ξέρουμε ότι η παρέμβαση των πολιτών σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατόν. Είναι κάτι που δεν μπορεί να διευθετηθεί στα γρήγορα. Πρέπει λοιπόν πραγματικά επίση να αξιολογούμε τον κίνδυνο χρεοκοπία. Στόχο τη έκθεση αυτή δεν είναι να δημιουργήσει ένα ταμείο, αλλά να φροντίσει το ταμείο αυτό να χρησιμοποιείται όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πώ χρησιμοποιώντα ένα μηχανισμό που υπάρχει σε άλλα ιδρύματα, ένα σύστημα peer review, ελέγχου δηλαδή μεταξύ ομοτήμων και να χρησιμοποιηθεί αυτό με ένα στάδιο αυτοαξιολόγησης. Υπάρχει στο Συμβούλιο της Ευρώπης αυτό το σύστημα για να αξιολογείται η ποιότητα της δουλειάς που γίνεται κατά της διαφθοράς και είναι κάτι που έχει δεχτεί η Ρωσία. Υπάρχει επίσης στον ΟΣΑ για την αξιολόγηση της δουλειάς που γίνεται για την ανάπτυξη και κατά της διαφθοράς και είναι κάτι που δέχονται όλες οι χώρες του ΟΣΑ. Και η Κίνα το δέχεται που είναι μέλος του ΓΚΑΦΙ. Άρα λοιπόν δεν είναι μηχανισμός που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, έχει δοκιμαστεί. Αφού λοιπόν χρησιμοποιείται για τη διαφθορά, μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί και για κάτι τόσο σοβαρό που είναι η χροκοπία των τραπεζών. Η ιδέα τώρα της ε, αυτοαξιολόγησης είναι πολύ σημαντική, γιατί θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μια τοπική τράπεζα κινείται. Πρώτα λοιπόν η αυτοαξιολόγηση. Μετά ο διάλογος και η συνεχής αμφισβήτηση των διαφόρων αρχών ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο. Υπάρχει έτσι μια ρουτίνα για να μην ξεχνάει ο καθένας τις ευθύνες του. Έχω υπόψη μου με την πρόταση αυτή ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Πρόκειται για την Ισλανδία, πώς κατέρευσαν εκεί οι τράπεζες. Ξέρετε ότι επηρεάστηκαν και χώρες της Ένωσης, οι οποίες είχαν θυγατρικές υποκαταστήματα Ισλανδικών τραπεζών, χωρίς να υπάρχει όμως έλεγχος και χωρίς να φροντίσουν να δούνε κατά πόσο υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος στην ίδια την Ισλανδία. 3,8 δισεκατομμύρια στήχησε στην Αγγλία, 600 εκατομμύρια στο Λουξεμβούργο, 800 εκατομμύρια στην Κεντρική Τράπεζα και όχι μόνο. ήτανε ε, μία αρχή ελέγχου που έπαιζε γκολφ με του υπουργού και με τους ε, τραπεζίτες. Αν υπήρχε το peer review, ο έλεγχος μεταξύ ομοτήμων, θα είχαμε δει το πρόβλημα νωρίτερα. Σίγουρα λάθη τεράστια πολλές φορές θα είχαν αποφευχθεί. Τέλος, πρέπει να περιορίσουμε τους κινδύνους. Εγώ βλέπω δύο πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, οι εποπτικές αρχές θα έπρεπε να φροντίζουν να περιορίζουν και να εμποδίζουν την μεταφορά των κερδών, των μερισμάτων και να διασφαλίζουν ότι είναι οι μέτοχοι και οι πιστωτές εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν τα πράγματα πριν να τα αναλάβει ο φορολογούμενος. Έπειτα, ο τραπεζικός φόρος για τη χρηματοδότηση ε, των ε, τραπεζικών προβλημάτων πρέπει να είναι κάτι που θα εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες και να προσαρμόζεται βάσει διαφόρων ε, κριτηρίων ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος αφαιρεγγιότητας. Με τέτοια μέτρα μπορούμε να έχουμε ένα καλό πλαίσιο το οποίο θα πετύχει το στόχο του. Να έχουν οι συστημικές τράπεζες τον ρόλο που πραγματικά τους έχει δώσει ο πολίτης και όχι να κάνουν ζημιά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με δυσκολίες στις πιο μεγάλες τράπεζες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω την Άστρι Λούμεν, τον Μπόμεν, Χάρκμαν, Βεκιφόρτ και τον εαυτό μου στον κατάλογο μιλητών. Δεν ξέρω αν θέλει κανένα άλλο. Φέω, σημειώνω. Άλλος κανείς. Και μετά ο εισηγητής. Λοιπόν, κλείνει ο κατάλογος ομιλητών. Άστριτ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά το σκιωδησηγητή μα και άλλους συναδέρφους θα είμαι σύντομη. Έχω όμως να πω κάτι για τις τροπολογίες που κατέθεσα εγώ και να υπογραμμίσω κάποια γενικότερα στοιχεία. Στη συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη φορά είχα υπογραμμίσει και χαίρομαι που άκουσα και συναδέρφους να μιλάνε για το ίδιο θέμα. Είχα υπογραμμίσει λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το θέμα της μεταφοράς μέσα σε μία ομάδα. Δεν είναι δυνατόν τα περιουσιακά στοιχεία των θηγατρικών και των υποκαταστημάτων να εξαφανίζονται από την μητρική σε περίπτωση κρίσης και οι πελάτες τελικά των θηγατρικών και των υποκατεστημάτων ε, να μην έχουν τίποτα στα χέρια τους. Έτσι και υπάρξει χρεοκοπία. Με διάφορες τροπολογίες προσπαθώ να διορθώσω αυτή την κατάσταση. Τη στηρίζω, εννοείται απόλυτα. Πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία των θηγατρικών και των υποκαταστημάτων να προστατεύονται. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ μέσα συμφωνούν γι' αυτό. Έρχομαι τώρα στην δομή επίλυσης των κρίσεων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνει μέσα στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τραπεζών, παρόλο που αυτό ελοχεύει διάφορους κινδύνους και δυσκολίες. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να δημιουργηθεί και μία ανεξάρτητη δομή η οποία θα είναι πιο αποτελεσματική και η οποία δεν ε, κινδυνεύει να επηρεαστεί από ίδια συμφέροντα. Ξέρω ότι πρώτη Επιτροπή, σίγουρα θα το συζητήσουμε, αλλά το σύνολο, έτσι όπως εγώ το καταλαβαίνω, εγώ δηλαδή είναι πιο συνεκτικό, στέκει καλύτερα και ελπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί. Τέλος, δεν έχω κάνει με ένα άμεσα πρόταση, αλλά θέλω να διευκρινίσω και να υπογραμμίσω ότι στηρίζω τις τροπολογίες οι οποίες θέτουν σε αμφισβήτηση τη διάκριση που γίνεται ανάμεσα στις συστημικές και μη συστημικές τράπεζες. Έχω ήδη εξηγήσει γιατί τα είπε και ο Σκιώδης εισηγητής μας, η διάκριση αυτή μπορεί να ξεκινάει από κάτι καλό, από μια καλή πρόθεση, αλλά ξέρετε ότι ο δρόμος για την κόλαση είναι γεμάτος καλές προθέσεις, όπως λέμε. Στην πράξη λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν θα λειτουργήσει, στοιχηματίζω. Θα έπρεπε καλύτερα, όπως το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, και όπως προτείνεται με διάφορες τροπολογίες για τις διασυνοριακές τράπεζες, ο Βρετανός συνάδελφος, νομίζω από το ECR, είπε ότι πρέπει να είμαστε ε, προσεκτικοί γιατί εδώ πέρα δεν βλέπουμε παρά την ουρά του σκύλου. Συνεπώς, έχοντας δει τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί για το πρόβλημα αυτό, ε, συμφωνώ κι εγώ να μην γίνεται διάκριση ανάμεσα στις συστημικές και μη συστημικές τράπεζες για τους λόγους που εξήγησαν οι προλαλήσαντες. Η συγγετριά μας πρέπει να έχει καταλάβει ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή αυτή εδώ για να εγκαταλείψουμε την ιδέα αυτής της διάκρισης. Είμαι σίγουρη με συμβαστικές τροπολογίες θα καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική λύση για όλους. ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριος Μπούμαν. Έχω μία ερώτηση προς τους φίλους και τις φίλες του ΕΛΚ, γιατί δεν καταλαβαίνω τη θέση τους σε σχέση με τις άλλες νομοθετικές πράξεις τις οποίες συζητούμε εδώ. Ίσως είναι δικό μου το πρόβλημα. Είναι τόσο υψηλού επίπεδου που δεν την κατανοώ. Γι' αυτό θέλω τη βοήθειά σας. Έχω λοιπόν σκεφτεί το εξής. Στις συζητήσεις αυτής της Επιτροπής έχει υπερισχύσει η εξής άποψη εξετάζοντας τον τραπεζικό τομέα και των χρηματοπιστωτικών ιδρωμάτων πίστευα ότι όλοι πιστεύουμε ότι η, η προσέγγιση ένα καλούπι ταιριάζει σε όλους είναι εσφαλμένη. One size fits all. Ότι αυτό είναι λάθος διότι διαφορετικά λειτουργούν, διαφορετικά ρίσκα αναλαμβάνουν και διαφορετικές ε, δραστηριότητες εκτελούν. Οι τράπεζες που λειτουργούν τοπικά και περιφερειακά εξυπηρετούν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν πρέπει αυτούς αυτά τα ιδρύματα να τα επιβαρύνουμε περισσότερο με ένα ακόμα πιο περίπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο. Αλλά θέλουμε να συγκεντρώσουμε όλες μας τις προσπάθειες σε αυτά τα ιδρύματα τα οποία αναλαμβάνουν αλλά και δημιουργούν τεράστιους κινδύνους. Και γι' αυτό ε, επιδιώξαμε ε, τον συμβιβασμό στην εποπτεία, στον τομέα της εποπτείας. Ο εισηγητής κ. Μαγκάλιο έκανε τον σωστό ορισμό και η ερώτηση της κυρίας Σβίνμπορμερ ε, ήταν σωστή ε, όσον αφορά τη διάκριση συστημικών ή μη συστημικών τραπεζών όταν μιλάμε για διασυνοριακές τράπεζες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε υπερατλαντικό επίπεδο. Είπαμε λοιπόν στην έκθεση του κυρίου Μαγκάλιο ότι δεν θέλουμε αυτό να το λύσουμε εξάντε, αλλά διαδικαστικά μέσω του Εποπτικού Συμβουλίου για τους Κινδύνους. Οπότε σωστά τέθηκε το ερώτημα, αλλά η απάντηση είναι πρόρη. Και κύριε Κάρας, όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια, την οδηγία για τα ίδια κεφάλαια, είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε μια σαφή, ε, ένα σαφή διαχωρισμό Εάν υπάρχει ένας φορέας ή ιδρύματα τα οποία έχει άμεση σχέση με τους πελάτες, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που μπορεί να ξέρει ποια προβλήματα έχει ο πελάτης, ο πελάτης ή εάν είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δεν έχει άμεση σχέση και επαφή με τους πελάτες και έχει, ας πούμε, ε, αναλαμβάνει άλλους κινδύνους αφηρημένης φύσης, δηλαδή πέραν των, προσωπικών συναλλαγών με τους πελάτες, επενδυτικούς κινδύνους, ιδιωτικές επενδύσεις κλπ. Τώρα όμως οι συνάδελφοι του ΕΛΚ συμπεριφέρονται τελείως αντίθετα. Αυτός λοιπόν ο διαχωρισμός στον οποίο είχαμε καταλήξει σε άλλες συζητήσεις άλλων νομοθετικών πράξεων δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να αντιστραφεί, δεν μπορούμε ξαφνικά να έχουμε 40 διαφορετικές προσεγγίσεις, διότι έτσι καταραίουν όλες μας οι αρχές, όλες μας οι κατευθυντήριες γραμμές επί των οποίων βασιστήκαμε, συζητήσαμε και για τις εποπτικές αρχές και στα CAD, όλα αυτά τα έχουμε πει και είπαμε ότι η Κομισιόν πρέπει να ασχοληθεί με όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διότι όλα κινδυνεύουν ή όλα είναι επικίνδυνα. Δεν το θεωρώ αυτό ούτε λογικό, ούτε, δεν είναι μια λογική προσέγγιση, ούτε ρεαλιστικό. Δεν είναι όλε, όλα τα ιδρύματα αυτά ίδια. Ευχαριστώ. Δεν ε, ξέρω αν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν ξέρω ακριβώς σε τι αναφερθήκατε. Όμως θέλω να εξηγήσω γιατί προτιμώ τη διατύπωση cross-border banks αντί για systemic banks. Το συστημικό ρίσκο, η συστημική τράπεζα ε, είναι τώρα μια ορολογία της μόδας, μια καραμέλα την οποία επιπλήζουμε με μεγάλη ευχαρίστηση, ενώ τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Οι τράπεζες στην Ισλανδία, ε, ναι, είχαν συστημικούς κινδύνου ε, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να ισχύει επειδή είχαν συναλλαγέ διαστηνοριακέ, Ε, αλλά μπορεί να λειτουργήσουν σε ένα ενδεχομένο συστημικό πλαίσιο. Δηλαδή είχαν διασυνοριακές συναλλαγές και γι' αυτό ήταν σε επικίνδυνη κατάσταση, αλλά ήταν συστημικέ. Ε, εάν κολλήσει την ετικέτα συστημική, τότε θα πεις ότι αυτή είναι μια τράπεζα η οποία δεν πρέπει ποτέ να κλείσει ποτέ να χρεοκοπήσει. Που σημαίνει ότι τελικά οι τράπεζες αυτές συνεχώς θα αυξάνουν το βαθμό του κινδύνου, όλοι θα, θα αναλαμβάνουν και χειρότερους κινδύνους, διότι ξέρουν ότι τελικά δεν θα, δεν θα επιτραπεί, δεν επιτρέπεται να χρεοκοπήσουν. Ενώ ε, αυτό, αυτό είναι αντιποραγωγικό ε, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι τράπεζες θα πρέπει κάποια στιγμή εφόσον λειτουργούν λάθος ε, και να μπορούν να κλείσουν, να, να χρεοκοπήσουν. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε με προσοχή το, το, το πλαίσιο λειτουργίας μας το οποίο μπορεί να δημιουργήσει συστημικά ρίσκα το πρόβλημα που είχαμε δεν ήταν η αφαιρεγγιότητα των τραπεζών τόσο πολύ όσο η έλλειψη ρευστότητας. Επίσης ε, αναγκάστηκαν να ξεπουλήσουν ε, στοιχεία του ενεργητικού το οποίο δημιούργησε πρόβλημα. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός όταν ε, ονομάζουμε τον, έναν κίνδυνο συστημικό. Δεν μπορούμε, πιστεύω, ποτέ να καθορίσουμε ακριβώς τι είναι συστημικό και τι δεν είναι. Απάντω στον κύριο Σμιτ για το Ταμείο. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με ένα καινούριο ταμείο. Σε λίγο θα υπάρχει ένα ταμείο για όλα τα προβλήματα. Ένα ταμείο για όλους και για όλα. δεν ε, νομίζω ότι θα, <laughs> θα καταλήξουμε σε ένα ταμείο για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ε, για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικέ κρίσεις πρέπει να έχουμε σταθερή οικονομική ανάπτυξη. Ε, αυτός πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος παρά να η δημιουργία συνεχώς νέων ταμείων. Ε, αυτό το λέω για να περιπλέξω ακόμα περισσότερο την ιστορία για τον κύριο Σμιτ. Το θέμα του ηθικού κινδυνού του moral hazard αυτό που βλέπουμε στο δικό μου κράτος μέλος είναι επειδή υπάρχει το Ταμείο Εγγύησης των Καταθέσεων, βλέπουμε νορμάλ ανθρώπους που παίρνουν τις καταθέσεις τους από καλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, των οποίων η διαχείριση έχει γίνει πάρα πολύ συνετά και να καταθέτουν σε άλλες τράπεζες οι οποίες ενεργούν επικίνδυνα απλώς και μόνο επειδή η κυβέρνηση έχει εγγυηθεί τις καταθέσεις. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός της προτάσεως. Δεν θέλουμε τα ταμιαυτήριά μας να γίνουν τελικά τράπεζες ανάληψης κινδύνων. Αλλά αυτός είναι ο λόγος, αυτό είναι το υπόβαθρο για τον οποίο οι καταθέτες μετακινούν τις καταθέσεις τους σε πιο επικίνδυνα ιδρύματα. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τους καταθέτες και τους πιο ευάλωτους, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε εν γνώση, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό το moral hazard, αυτό το, θέμα υπάρχει, είναι πραγματικότητα. Ε, δεν έχω αντίρρηση να προσθέσουμε ένα-δύο ακόμα εργαλεία στο βαλιτσάκι των εργαλείων, στο toolbox, Ορισμένα από αυτά τα μέσα, τα εργαλεία μπορεί να είναι πάρα πολύ λογικά. Γιατί λοιπόν όχι. Γιατί να μην το συμπληρώσουμε. Μου άρεσε η πρότασή σας που λέει ότι η ρυθμιστική αρχή θα πει στην τράπεζα δεν μπορείς να αλλάξεις το μοντέλο, το μοντέλο λειτουργίας σου, παραδείγματος χάρη, και να χρησιμοποιήσεις κάτι άλλο. αντί παραδείγματος χάρη να γίνεται συνεχώς η μετατροπή χρέους σε μετοχές, σε μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης, η δυνατότητα του, της ρυθμιστικής αρχής να ελέγξει ενδοετερικές μεταφορές των ε, στοιχείων του ενεργητικού. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδίω αν έχουν γίνει πριν από την ε, χρεοκοπία. Τι, τις είδους μεταφορέ ε, ε, μεταφορές του ενεργητικού έχουν γίνει πριν, πρόσφατα, δηλαδή πριν, πριν δηλωθεί χρεοκοπία. Εκεί πρέπει να μπορούμε να εφαρμόσουμε μέτρα διαφάνειας για να ελέγξουμε αυτήν την διαφυγή κεφαλαίων. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ορισμένες τράπεζες έχουν επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία λειτουργούν πάρα πολύ καλά ε, επί τη βάση κεφαλαϊκών, ε, καλά οργανωμένων κεφαλαϊκών ε, θυγατρικών. Δεν είναι λοιπόν απλό να πούμε ότι ε, παίρνουμε όλα τα χρήματα πίσω και ε, χειριζόμαστε όλους τους εμπλεκόμενους με τον ίδιο τρόπο, ισότιμα. Ε, μην ξεχνάμε ότι ορισμένε από αυτές τις μεγάλες τράπεζες που είχαν επιτυχείς σιγατρικές λειτουργούσαν ένα πολύ επιτυχημένο λειτουργικό μοντέλο. Εάν τιμωρήσουμε Α, εάν θέλουμε οπωσδήποτε να καθορίσουμε ποιες είναι συστημικές ε, τράπεζες, σίγουρα θα μας ξεφύγουν μερικές. Δεν μπορούμε, πιστεύω, να ε, ορίσουμε συστημικές ε, τράπεζες, τις τράπεζες που έχουν διασυνοριακές συναλλαγές. Ακόμα και στη δική μου χώρα, ορισμένες μικρές τοπικές τράπεζες απέτυχε, χρεοκόπησαν. Ε, και σε άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει σωστή εποπτεία των μικρών τραπεζών και σε τοπικό επίπεδο, διότι διαφορετικά μπορεί και αυτές να γίνουν συστημικές. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ο όρος συστημικό, systemic banks είναι ο καλύτερος, cross-border πιστεύω, διασυνοριακές είναι ο καλύτερος όρος για να χρησιμοποιήσουμε για το ψήφισμα. Ο κύριος Φέο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για τη σοβαρή δουλειά που μας παρουσίασε. Δεν θα ήθελα να μπω στο θέμα των ορισμών όσον αφορά τη διασυνορική τράπεζα, τη συστημική τράπεζα. Θέλω απλώ να πω το εξή. Εδώ ασχολούμαστε με θέματα που μπορεί να έχουν νομοθετικέ συνέπειε. Και εφόσον λοιπόν έχουν νομοθετικέ ε, συνέπειε, η ομοιομορφία των ενιών που χρησιμοποιούμε στα διάφορά μα ε, μέσα είναι πολύ σημαντική. Εάν καταφέρουμε με αυτή την ομοιομορφία εφαρμογής, να φτάσουμε σε μια λύση λογική, το καλύτερο είναι να χρησιμοποιούμε πάντοτε ομοιόμορφες έννοιες και ορισμούς. Εν τέλει, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή που έχει σχέση με το early intervention, την ε, έγκυρη παρέμβαση. Αυτό έχει να κάνει με την δημοσιοποίηση της παρέμβασης. Υπάρχουν τράπεζες οι οποίες ανησυχούν σε σχέση με αυτό το ίδιο θέμα. Θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνει δημοσιότητα το γεγονός ότι ένας επόπτης παρεμβαίνει σε μια προκαταρτική φάση. Γιατί αν αυτή η παρέμβαση πάρει δημοσιότητα θα έχει συνέπειες στην αγορά που μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν σε σχέση με, μια, με την εμπιστοσύνη σε ένα συγκεκριμένο μόνο θεσμό η χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Και ήθελα να επιστήσω την προσοχή της εισηγήτριας σε αυτό το θέμα για να μπορέσει να μας καθησυχάσει. Ευχαριστώ. Ζητάω το λόγο και ευχαριστώ, παρόλο που είχε κλείσει ο κατάλογος ομιλητών, για να απαντήσω σε αυτά που ακούσαμε πριν. Ευχαριστώ και εγώ βέβαια την Ελίζα. Λοιπόν, κοιτάξτε, σε αυτό το στάδιο πρέπει να παραδεχτούμε ότι ψάχνουμε τις καλές έννοιες. Και αυτά που είπε Ούντο, ότι δεν υπάρχει συνοχή, πολύ θεμητό, αλλά είναι φυσιολογικό. Σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε, να σκεφτούμε, να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες. Συμφωνώ και με τη Βίκη. Σπάνιο, ε? γι' αυτό και το υπογραμμίζω. Είναι αλήθεια ότι τα δύο κριτήρια τα οποία είναι να έχουμε ένα κατάλογο συστημικών ιδρυμάτων ή να πούμε διασυνοριακά, δεν φτάνουν. Και μάλιστα για την Ευρωπαϊκή Έκθεση, για την έκθεση μάλλον για την Ευρωπαϊκή Αρχή Συστημική, προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Στην εσωτερική αγορά υπάρχει ένα σοβαρός λόγος και εξαιτία του μεγέθους τους που είναι ένα από τα κριτήρια, όχι το μόνο, για τον οποίο είναι συστημικές ε, οι αυτές αυτέ ομάδε, αλλά μπορεί, όπω είπε και η Βίκη, να υπάρχουν και μικρά ιδρύματα ή προϊόντα τα οποία χειρίζονται κάποιες ε, τράπεζες και που να μπαίνουν σε αυτή την κατηγορία. Και γι' αυτό και υποβάλαμε τις τροπολογίες μα. Δεν είναι σε αντιπαράθεση. Πρέπει να καλύψουμε όλες τι περιπτώσει χωρί απριόρι, χωρίς να κάνουμε διάκριση λόγω ιδεολογία. Όντω, όταν πρόκειται για διασυνοριακά ιδρύματα, υπάρχει ο κίνδυνο ε, να μεταφερθούν τα προβλήματα από τη μέση στην άλλη χώρα. Υπάρχει τώρα η Επιτροπή Κινδύνου. Το όργανο αυτό πρέπει να μπορεί να αναπτύξει τα κριτήρια. Μα γι' αυτό υπάρχει. Το δημιουργούμε το όργανο αυτό γιατί πιστεύουμε ότι προς το παρόν δεν έχουμε δουλέψει αρκετά πάνω στα κριτήρια που μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε εκ των πριτέρων έναν κίνδυνο. Να πούμε ότι εδώ υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε κίνδυνο. Συμφωνεί φαντάζομαι και η Ελίζα για το ότι δεν πρέπει να μονοπολούμε στη μία κατηγορία στην άλλη τους κινδύνους. Με αυτά που έχουν αποφασιστεί ή που θα αποφασιστούν με το πακέτο εποπτείας που έχετε ψηφίσει εδώ στην Επιτροπή αυτή, να συνεχίσουμε αφήνοντας ανοιχτό. Τώρα ο κύριος Μπούμαν μόλις τώρα ήρθε, για εκείνον τα έλεγα όλα αυτά. Δεν μου άκουσε τι να κάνουμε. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Εγώ είμαι η τελευταία ομιλήτρια για αυτό το θέμα. Μετά η συγγήτρια πάλι θα πάρει το λόγο. Έχω και εγώ να πω μερικά πραγματάκια. Και εμένα αυτό με απασχολεί. Έχω την τροπολογία 140 εξάλλου που λέει και συστημικά και διασυνοριακά ιδρύματα. Έβαλα και τα δύο. Γιατί και εμένα με απασχολεί αυτό το θέμα. Γιατί η Λίμαν μπορεί να είναι συστημική και σε μια χώρα που δεν βρισκόταν. Και μπορεί να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Και εδώ επανέρχομαι λιγάκι στο θέμα της εσωτερικής αγοράς. Γιατί εμένα με απασχολεί πολύ. Σε μια εσωτερική αγορά που δεν έχουμε όσον αφορά την φερεγκιότητα. ιδιαίτερα στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ιδρυμάτων, ξέρουμε ότι αν κάτι πάει στραβά, οι επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές. Και με τη Solvency 2 το βλέπω αυτό πιο έντονα. Τώρα έρχομαι στη φύση του ταμείου. Εγώ δεν αγαπάω εξορισμού τα διάφορα ταμεία, αλλά αυτό το ταμείο, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, τελικά είναι ένα μικρό ταμείο που χρησιμοποιείται προκειμένου να παρεμβαίνει στην περίπτωση επίλυσης ή διαχωρισμού ξέροντας τι πρέπει να κρατήσουμε, συστήματα πληρωμής για παράδειγμα, τα διαχωρίζουμε από άλλα πράγματα. Δεν είναι ένα ταμείο για να πληρώνει διαφέρει από τον deposit guarantee, με εγγύηση καταθέσεων. Δεν δημιουργεί τους ίδιους κινδύνους. Δεν είναι bailout. Εσείς Αν δηλαδή ένα ίδρυμα φτάσει σε κάποια μεταρρύθμιση με κάποιες, ε, κάποια πρόστιμα, πληρωμές και αρχίζουν να δημιουργούνται ένα σωρό άλλα προβλήματα, δεν είναι bailout αυτό το ταμείο. Είναι ένα μέσον για να έχουμε θεμητή, δίκαια, σύμφωνα με τους κανόνες, δηλαδή μεταφορά ενεργητικού από τη μία πλευρά στην άλλη. Οι επόπτες μπορεί να πούν ότι αυτό το κεφάλαιο νίκη στην Πολωνία, ναι, αλλά στέλνει χρήματα σε μια άλλη χώρα και εκεί παρεμβαίνουν οι επόπτες. Για το ομένο Βασίλειο ισχύει η περίπτωση των ε, μεταφορών μέσω Ατλαντικού. Περίπτωση Λίμαν. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα μέσο το οποίο να επιτρέπει ...αυτή τη σωστή κατανομή πόρων με fair play, δίκαια, εκεί όπου πρέπει να πάνε, εκεί όπου ανήκουν. Εγώ έτσι το βλέπω. Αυτό σημαίνει group transfers για μένα. Δεν θα πρόκειται για φέρετες αποφάσεις, πρέπει να εντάσσονται στο γενικότερο σύστημα και να καθορίσονται από πριν το πώς θα γίνονται. Πρέπει από πριν να ξέρουμε αυτή η επίλυση πώς θα γίνεται. Και η εποπτεία θα πρέπει να εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η επίλυση της κρίσης, η διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης. Σε αυτή την περίπτωση η δίκαιη κατανομή δεν αποτελεί εμπόδιο. Επίτηδες χρησιμοποιούμε το burden sharing, αλλά προσοχή. Εδώ πρόκειται για ένα ταμείο που έχει φτιαχτεί, υπάρχει και χρησιμοποιείται βάσει προκαθορισμένων κανόνων, ανάλογα με τις ανάγκες. Δεν είναι burden sharing, δεν είναι κατανομή βάρους όπως συνήθως το αντιλαμβανόμαστε στο πλαίσιο του bailout. Δεν είναι αυτό. Και επειδή οι επόπτες πρέπει να μπορούν να επηρεάζουν τα πράγματα, το είπα και στην διάσκεψη που ήμουνα με τον Επίτροπο, είναι πολύ σημαντικό οι επόπτες, οι τραπεζικές αρχές να έχουν κάποια, κάποιους ειδικού ε, για την αφαιρεγκαιότητα για να μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο έχει γίνει, γίνεται η διαχείριση της επίλυσης με το σωστό τρόπο, η διαχείριση της κρίσης με το σωστό τρόπο. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια ομάδα, μια ενότητα μέσα στην τράπεζα που να ασχολείται με την διαχείριση της κρίσης. Ελπίζω να υπάρχει και αυτή η πραγματογνωμοσύνη για την αφαιρεγκιότητα. Οι προτάσεις πάντως έγιναν από τον Επίτροπο Μπαρνιέ και εγώ αυτό που κατάλαβα τότε ήταν το Ταμείο Μπαρνιέ θα χειριζόταν 50 με 70 δις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από τη Γερμανία μίλησαν για ένα δισεκατομμύριο το χρόνο από τις τραπεζικές εισφορές. τότε όμως δεν παίρνετε μεγάλα ποσά από τις άλλες εισφορές ή φόρους που θέλετε να φτιάξετε. Το άλλο επιχείρημα που έχει χρησιμοποιηθεί για την πρόταση Μπαρνιέ είναι ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να χρησιμοποιούν ό,τι μπορούν για να πληρώσουν τα ελλείμματα. Τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει όμως ένα τέτοιο ταμείο εφόσον έχει φτιαχτεί καλά να ασχολείται με το ενεργετικό του ισολογισμού στη Σουηδία για παράδειγμα και από ό,τι κατάλαβα τα είδαν όλα αυτά με λεπτομέρειες και εγώ προσπάθησα να έχω μια ανταλλαγή απόψε και με τη Eurostat πώς έχουν τα πράγματα. Το μοντέλο Μπαρνιέ έχει να κάνει περισσότερο με το εθνικό επίπεδο, όχι τόσο με το ευρωπαϊκό. Εμείς πάντως με την έκθεση Μαρσία Μαργάγιο το έχουμε βάλει σαν Ευρωπαϊκό Ταμείο. Ίσως μπορούμε να τα συνδυάσουμε τα δύο σε ένα σύστημα. κάποια στιγμή ίσως πρέπει να το δεχτούμε αντί να βάζουμε βέτο εδώ που έχουμε φτάσει. Να πρέπει να υπάρχει δηλαδή και ένα εθνικό στοιχείο. Να λέμε είναι στον ισολογισμό και λειτουργεί σαν δίκτυο ασφαλείας, σαν δίκτυ. Δεν ξέρω βέβαια οι συνάδελφοι πώς το βλέπουν. Ίσως μπορούμε όμως να βοηθηθούμε και για το εποπτικό πακέτο. Αυτά είχα να πω. Και συγγνώμη, λέει προς την εισηγήτρια πρόεδρος, που δεν μπόρεσα να έρθω νωρίτερα να σας δω τέτα τέτ και να τα πω όλα αυτά και τα λέω τώρα. Ελίσα. Η εισηγήτρια γιατί εγώ ήμουν η τελευταία στον κατάλογο μιλητών. Ελίσα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μου είπατε. Όλα μου φάνηκαν πολύ σημαντικά και μας επιτρέπουν να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό. Κανένας δεν είναι απόλυτα σίγουρος για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Πέρα από ιδεολογικές διαφορές, το θέμα είναι πώς θα το λύσουμε. θα αναφερθώ σε θέματα και όχι στις παρεμβάσεις του ενός και του άλλου. Λοιπόν, ένα πολύ ζωτική σημασία θέμα είναι το με ποιο χώρο ασχολούμαστε. Το ευρωπαϊκό καθεστώς. Για ποιο πράγμα ακριβώ, για ποιο χώρο μιλάμε. Είναι το ίδιο με αυτό που είχαμε πριν από δύο-τρει εβδομάδε όταν συζητήσαμε την έκθεση Μαργάγιο και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί τα επιχειρήματα υπέρ μιας πλήρους κάλυψης των διασυνοριακών συναλλαγών, και ορισμένοι το είπανε, είναι αδύνατον στην πράξη. Πρέπει να δούμε την ευρωπαϊκή διάσταση καλύτερα, γιατί αλλιώς η εποπτική αρχή, το EBA, αρχίζει να ελέγχει όλες τις διασυνοριακές τράπεζες, κάτι το οποίο δεν χρειάζεται, θα γίνει γραφειοκρατία. Οπότε η συνένεση στην οποία φτάσαμε νωρίτερα είναι ακριβώς αυτό που ανέφεραν και Σίλβια και άλλοι. Θέλουμε να καλύψουμε τράπεζες και όλοι Σμιτ αυτό είπε 50-40 διασυνοριακές τράπεζες και οι τράπεζες λένε ναι να εντοπιστούν. Θα είναι η υπηρεσία η οποία θα ταξινομήσει και θα πει γιατί κινδύνους μιλάμε. Εντάξει, δεν είναι μόνο το μέγεθος, το μέγεθος είναι ένα κριτήριο, αλλά και το πόσο πολύπλοκη είναι η διαχείριση, κατά πόσο υπάρχει έλλειψη διαφάνειας, υπάρχουν και άλλα στοιχεία δηλαδή εκτός από το μέγεθος. Μια από τις κύριες πτυχές, συνεπώς, που πρέπει να κατανοήσουμε και πάνω στην οποία πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι αν κρατήσουμε την συνένεση, για το για ποιο πράγμα μιλάμε, ποιο είναι το πεδίο μας. Εφόσον συμφωνήσαμε για την έκθεση Μαργκάγιο, νομίζω ότι πρέπει να είναι το ίδιο. Και εγώ στις προσεβαστικές μου τροπολογίες τι έκανα. Συμπεριέλαβα αυτή την ιδέα γιατί εγώ κατάλαβα ότι αυτό ήθελε το Κοινοβούλιο και αυτό ήθελε η Επιτροπή μας. Το ίδιο δηλαδή το οποίο συμφωνήσαμε πριν από δύο εβδομάδες εδώ στην Οικονομική Επιτροπή. Και συζήτησα με την Τανούδα Χούμπνερ και με τους άλλους σκιώδε που ήταν ε, παρόντες και αυτό κατάλαβα, όπως και Ούντο και Σιλβί και ο Φέο και άλλοι. Το ζήτημα είναι, συνεχίζουμε στην ίδια γραμμή, συμφωνούμε, αλλιώς καταραίει το όλο οικοδόμημα. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει αυτό το ΕΛΚΑ και να συμφωνήσει με αυτά που έχουν προαποφασιστεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Για τα άλλα τώρα. Για το toolbox. Εγώ έχω συμπεριλάβει στις προσεβαστικές μου τροπολογίες όλα τα σχετικά στοιχεία. Γιατί τα περισσότερα από αυτά, περίπου όλα, είναι μια προσθεθέμενη αξία για το κείμενο προσπαθούσα να δώσω παραδείγματα για κάποιες πολύ λεπτομερές τροπολογίες, αλλά δεν νομίζω ότι αυτές είναι οι τροπολογίες που πρότειναν όσοι πήραν το λόγο εδώ. Το Toolbox λοιπόν είναι μια επιτυχία. Τώρα, ένα δεύτερο θέμα. Η κυρία Λούλινγκ αναφέρθηκε σε αυτό και νομίζω ότι και η Ντανούντα Χούμπνερ μέσω του κύριου Κάρα το έθεσε κι άλλοι. Όλες οι τροπολογίες που πάνε προς την ίδια κατεύθυνση πρέπει όντως να εγκρεθούν. Και ελπίζω ότι η συμβαστική μου πρόταση θα καλύψει αυτό που θέλετε. Ο κύριος Σφαίο επίσης ανέφερε κάτι σημαντικό, το θέμα του απόρριτου σχετικά με το τι κάνουν οι υπόπτε. Υπήρξε μια τροπολογία για το απόρριτο από τη Σιλβί Γκουλάρ που πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Εννοείται ότι αυτό είναι μέρος της δουλειάς της εποπτικής αρχής, της CBA. Εννοείται, ποτέ δεν πρέπει να έχουμε δημόσια συζήτηση. Αν θέλει κάποιος να παρέμβει, να συζητήσει, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι δείκτες της EBA soft triggers με hard triggers. Για το ρόλο των ταμείων. Αυτά που είπε η Sharon εδώ στο τέλος καλύπτει λίγο πολύ αυτό που ήθελα και εγώ να πω. Αν πάμε σε εθνικά ταμεία, ακόμα κι αν αυτό είναι ο συμβιβασμός, δεν πρέπει να αφήσουμε απ' έξω την ευρωπαϊκή διάσταση γιατί αλλιώς κατακαιρματίζουμε την εσωτερική αγορά σε κομματάκια. Ο ρόλος του EBA ή του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου είναι ότι ακριβώς υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση και εφόσον πρέπει να έχουμε συμβασμό μην το χάσουμε αυτό το στοιχείο. Ή που θα ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά ή θα τη χάσουμε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να το προστατεύσουμε. Πέρα από αυτά τώρα, μεθοδολογικά, προτείνω την επόμενη εβδομάδα να οργανώσω τους τελικούς συμβιβασμούς και να τους συζητήσουμε τη βδομάδα του Στρασβούργου. Έτσι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια αμοιβαία κατανόηση, να ξέρουμε δηλαδή τι θα ψηφίσουμε, τι ακριβώς θέλουμε. Και μετά με τους συνεργάτες μου και τους συνεργάτες σας θα στείλω κάποιες συμβαστικές προτάσεις για να δω κατά πόσο καλύπτουν τους ε, στόχους σας. Αυτά δηλαδή που είπατε σήμερα. Πάντως, θεωρώ ότι το ΕΛΚΑ συνεχίζει να συμφωνεί με αυτό που αποφασίσαμε για το πεδίο εφαρμογής. Γιατί είναι κάτι ουσιώδες και που πρέπει έτσι κι να είναι προκαθορισμένο αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Αλλιώς θα είμαστε σε κινούμενη άμμο και δεν είναι ότι καλύτερο για να κάνουμε διαπραγματεύσεις σε τέτοια βάση με τα άλλα κοινωτικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλους σας για τις παρεμβάσεις σας και ελπίζω οι συμβαστικές μου προτάσεις να καλύψουν όλες τις ανησυχίες όσων πήραν το λόγο εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εγώ Ελίζα 22 Ιουνίου θα ψηφιστεί για... και μετά θα πάει στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Προχωρούμε στο θέμα 17 ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Εισηγητής ο κύριος Κάρας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ καταρχάς τους, ο, τους κοιόδης εισηγητές με τους οποίους συνεργάστηκα θαυμάσια έχει περάσει η ώρα ε, και έχω να σας πω το εξής. Ήδη σημειώσαμε μια πρώτη επιτυχία. ο οποίο απαιτεί όμως ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από μας. Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου συμφώνησε με την ομάδα της Eurostat και την ερχόμενη εβδομάδα στο ΕΚΟΦΗΝ θα, θα συζητηθεί ως σημείο α η προτινόμενη ρύθμιση της Eurostat. Ξέρω ότι όσο το, τόσο το Συμβούλιο όσο και η Eurostat συμφωνεί με το ε, έχουν μάλλον επιχειρηματολογήσει κατά του πνεύματος και της δικής μου έκθεσης αλλά και των συζητήσεων που είχα κάνει εγώ με το Συμβούλιο. Και ξέρω ότι και το Συμβούλιο και η Eurostat έχουν πει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να θεωρήσει, ε, ε, ε, θεωρεί την πρόταση της Κομισιόν ως ελάχιστο, ελάχιστη πρόταση, ελάχιστες απαιτήσεις και ότι θέλει να διευρύνει την πρόταση της Κομισιόν ενώ ε, πολλά από τα σημεία τα οποία είχαμε εμείς προτείνει ήδη έχουν συμφωνηθεί, τα, έχουν περάσει από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ και είναι πολύ ευχάριστο. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε γρήγορα και οργανωμένα. Προτείνω ήδη τον Ιούνιο να ψηφίσουμε στο Κοινοβούλιο το ψήφισμα ε, και την προφορική ερώτηση στο, στην Ολομέλεια, συγγνώμη, και τον Ιούλιο να ψηφίσουμε την νομοθετική ε, πράξη. Για να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να δώσουμε το πολιτικό μήνυμα της βούλησης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό σας παρακαλώ την νομοθετική γνωμοδότηση, το ψήφισμα, προφορική ερώτηση, να καθορίσετε έτσι το χρονοδιάγραμμα ώστε μαζί να αποφασίσουμε τον Ιούνιο προφορική ερώτηση και ψήφισμα και το αργότερο τον Ιούλιο την νομοθετική πράξη. Δεύτερη παρατήρηση. Ανεξάρτητα από την συμφωνία εντός του Συμβουλίου και το, το ότι επιτεύχθη επειδή εμείς ασκήσαμε έντονη πίεση δεν σημαίνει και ότι θα ολοκληρωθεί όλο το νομοθετικό έργο σωστά, όπως το επιθυμούμε. Προς το παρόν τα πράγματα έχουν εξελιχθεί όπως θέλαμε εμείς. Ε, εμείς ζητήσαμε από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου να εξετάσει το ενδεχόμενο της εφαρμογής της διαδικασίας συναπόφασης βάσει του άρθρου 126 που θα αποτελεί την νομική βάση. Στη νομική βάση όμως τα στατιστικά είμαστε μέσα στη συναπόφαση. Ε, για μένα δεν πρόκειται για θεσμικό πρόβλημα, αλλά το ερώτημα είναι να διασφαλίσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου εκεί όπου πρέπει να παίξει ένα ρόλο. Δεδομένου ότι εμείς εδώ πολεμάμε να βελτιωθεί η πρόταση της Κομισιόν. Άρα λοιπόν θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Κομισιόν μέσα στη συναπόφαση. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε, ε, ε, αν μπορούμε να το κάνουμε. Μέχρι τώρα ενήργησα και συνέταξα την έκθεσή μου έτσι, ως, σαν να βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία της συναπόφασης η διαδικασία δεν θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά θέλουμε αυτή τη διευκρίνηση. Είμαστε στην, συναπόφαση ή δεν είμαστε. Και τέλος πρέπει να ενεργήσουμε πολιτικά, διότι για μένα το ερώτημα της ε, ε, Eurostat και του ρόλου της Eurostat είναι το η πρώτη νομοθετική πράξη η οποία προκύπτει από τις εμπειρίες που είχαμε με την Ελλάδα. Και είναι πραγματικά η ώρα της αλήθειας για να δούμε εάν τα παθήματά μας γίνανε μαθήματα και αν είμαστε σοβαροί στο να θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχου. Πρέπει λοιπόν να μείνουμε στις θέσεις μας, να είμαστε συνεπείς και να ολοκληρώσουμε το συνεπές νομοθετικό έργο. Γι' αυτό ακριβώς και κάναμε το διαχωρισμό ε, αφενός ψήφισμα, αφετέρου προφορική ερώτηση και συνεχεία νομοθετική πράξη. Δηλαδή δίνουμε ένα πολιτικό μήνυμα και εκφράζουμε τη βούλησή μας. Με τους κοιόδης εισηγητές ε, συζήτησα τις ε, προτάσεις ε, και ε, βεβαίως θα συζητήσουμε όλες τις καλές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι καλές. Και όλα τα μέτρα τα οποία ζητήσαμε να εφαρμοστούν από το 2004 μέχρι το 2007 πρόταση Αλμούνια, έκθεση ΣΒΑΠ, η δική μου έκθεση του 2005, ε, συντονισμός με τις ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, μηχανισμοί κυρώσεων. Όλα αυτά τα μέτρα που ζητήσαμε και δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί, υλοποιήσει να τα προχωρήσουμε. Για εμείς θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι η Eurostat πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα, ολοκληρωμένα Πλήρω δηλαδή, χωρίς κάθε φορά που θέλει να κάνει έναν έλεγχο ή να παρέμβει να χρειάζεται άδεια από τα κράτη-μέλη. Όταν θεωρεί ότι οι πράξει της και οι ενέργειέ της είναι σωστές, να μην συναντά κανένα πρόσκομα, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει τις ευθύνες της. Είναι υπεύθυνη η Eurostat και είναι ευθύνη της να έχει τα στατιστικά στοιχεία μέσω συνεργασίας, μέσω ενημέρωσης αλλά όχι να παίρνει κάθε φορά μία των προτέρων άδεια λειτουργίας ή εξάσκησης των δραστηριοτήτων της. Η Eurostat είναι ένα υπεύθυνο όργανο, πρέπει να είναι ελεύθερο να ενεργεί έτσι όπως νομίζει. Πρέπει να είναι ελεύθερη ε, και ανεξάρτητη, να μπορεί να συνεργάζεται με την Κεντρική Τράπεζα, να διενεργεί, να ε, εκτελεί επισκέψεις, αποστολές ελέγχου και ενημέρωσης. Όλα αυτά τα υποστηρίζουμε. Πιστεύω και το θεωρώ ως προϋπόθεση τον, ε, στην Ολομέλεια του Ιουνίου μπλοκ να μπορέσουμε να υπερψηφίσουμε το ψήφισμα διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό προσπάθησα εκ των προτέρων να συμφωνήσω με τους κοιόδης εισηγητές και τους είχα δώσει και το, το σχέδιο, το γνωμοδότησή μου σε μεταφρασμένη. Ευχαριστώ. Uh, thank you. Um, Ευχαριστώ. Ο πρώτος εισηγητής είναι ο κ. Σιτούνα, Έντουαρτ Σιτούνα, αν θέλει να μιλήσει. Ναι, θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω απολύτως τον κύριο Κάρας και την προσέγγιση του και την ε, πίεση που πρέπει να ασκήσουμε για να επιταχύνουμε την πρόοδο και να ολοκληρωθεί αυτή, να αναπεράσει αυτή η νομοθετική πράξη. Επίσης ε, θέλουμε η Eurostat να έχει την εντολή την οποία ζητάμε τώρα. Πιστεύαμε ότι είχε την εντολή και, και ήταν μεγάλο σοκ για μας να διαπιστώσουμε ότι η Eurostat δεν είχε την εντολή να εκτελέσει αυτά τα οποία θέλουμε. Θέλουμε λοιπόν το ταχύτερο να ξεκαθαρίσει, ξεκαθαριστεί το θέμα της εντολής ε, της Eurostat, να δοθεί αυτή η εντολή. Δεν έχω πρόβλημα με το ψήφισμα, ούτε με τις τροπολογίες. Είναι αρκετά ευρείες Επίσης συμφωνώ ότι κανένας έλεγχος από πλευράς Eurostat δεν πρέπει να έχει εμπόδια ή να προσκόμματα. Η μόνη μου παρατήρηση είναι ότι θα πρέπει να μην υπάρχει κανένα πρόσκομα ως προς τους φορείς ή τα πρόσωπα με τα οποία θέλουν να συζητήσουν οι εκπρόσωποι της Eurostat. Δηλαδή να μην εμποδιστούν σε καμία περίπτωση να συζητήσουν ή να διενεργήσουν συναντήσεις με υπουργεία, με ιδρύματα δημόσια, με πανεπιστήμια ή με άτομα. Δηλαδή να είναι ελεύθεροι στην προσέγγιση τους προς τα ιδρύματα ή τους φορείς που θεωρούν ότι πρέπει να προσεγγίσουν. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. απρόσκοπτη, απρόσκοπτη προσέγγιση, να έχει δηλαδή μια απρόσκοπτη ξεκάθαρη εντολή η Eurostat να μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε φορέα θεωρεί ε, αναγκαίο. Και εύχομαι ε, να ολοκληρωθεί επιτυχώς όλη αυτή η προσπάθεια στον εισηγητή. Ο Όλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αυτό το είδος τα θέματα που αφορούν στατιστικές δεν είναι και τόσο γοητευτικά ούτε σημαντικά από πολιτικής άποψης. Παλαιότερα δεν ήταν. Σήμερα όμως πιστεύω πως αν ρωτούσαμε το κοινό τι τους ενδιαφέρει, τον κόσμο στις χώρες μας, θα... είμαι σίγουρος ότι θα έλεγαν ότι δεν θα πρέπει κανεί να δίνει ψευδείς σε στατιστικές όταν είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά αυτό βρίσκεται πλέον πολύ ψηλά στην πολιτική ημερήσια διάταξη και πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα. Ο κύριος Κάρας πιστεύω έκανε πολύ καλή δουλειά και τον υποστηρίζω πλήρω καθώ και ο κύριο ε, Σικλούνα, όπως και ο κύριος Σικλούνα. Ίσως ε, θα έπρεπε ωστόσο να έχουμε κάποιες λεπτομέρειες και Νόμιζα ότι θα τις, προτείνατε. Όταν οι αρχές ε, του ανταγωνισμού μεταβαίνουν στις διάφορες χώρες δεν προειδοποιούν. Όχι, κάνουν ευνίδιους ελέγχους ε, και λένε ότι ορμούν μέσα, ανοίγουν την πόρτα και λένε να είμαστε. Εσεί ε, ναι και κουνάτε έτσι το κεφάλι σας συγκαταβατικά αλλά κανονικά είστε πολύ σκληροί κι εσείς. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνονται τέτοιου είδου ευνίδιε επιθεωρήσεις ή τουλάχιστον υπάρχει δυνατότητα για τέτοιες επιθεωρήσεις γιατί πολλές φορές ο φόβος ε, λειτουργεί αποτρεπτικά. Επίσης αναφέρεται εδώ το προσωπικό και ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε κάπως πιο ακριβείς σε σχέση με την ανάγκη να εξετάσουμε ίσως κάπως ε, πιο σφιχτή στον προϋπολογισμό. Νομίζω πως ε, θα μπορούσαμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε κάποιο δημιουργικό λογιστικό πρότυπο και αυτό εξαρτάται από την επιδεξιότητα του προσωπικού, την επιδεξιότητα των όσων προσπαθούν να είναι πολύ δημιουργικοί. Και αυτό είναι πάντοτε πρόβλημα. Το έχουμε δει ότι είναι πρόβλημα κάτι τέτοιο. Και ίσως να πρέπει και αυτό να το τονίσουμε. Κάτι ακόμα κύριε Πρόεδρε. μπορούσαμε να μιλήσουμε και για κυρώσεις. Κυρώσεις ε, στον τομέα αυτό, όχι σε ευρύτερο πλαίσιο, αλλά και όσον αφορά την ε, απόδοση λογαριασμών και τα σωστά στοιχεία σε σχέση με τις στατιστικές. Νομίζω πως γενικά συμφωνούμε, να είμαστε δηλαδή όσο γίνεται πιο σκληροί και αυστηροί. Ευχαριστώ. Μάλιστα, προσπαθείς ε, όλα να κάνεις τις στατιστικές πιο γοητευτικές με κυρώσεις και ευνίδιους ελέγχους. Ναι. Ε, ευχαριστώ η Κέι τώρα. Η Κέι ε, μιλώ εξ ονόματος και του συναδέλφου Φόξ. Είναι στην Επιτροπή Προπολογισμού για μια σημαντική ψηφοφορία. Θέλω ωστόσο να ευχαριστήσει τον εισηγητή για τη συνεργασία του και για όλη τη δουλειά που έκανε πριν να υποβάλει το σχέδιο έκθεσή του και γιατί ήταν πολύ ανοιχτό και συμπεριέλαβε τις ιδέες αυτές μαζί με τους ε, σκεώδεις. Ως μπορώ να υποστηρίξω το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Κάρας και να ε, καθώς συμπεριλαμβάνοντας αυτή τη γνωμοδότηση, ε, συμπεριλαμβάνει σε αυτή τη γνωμοδότηση ιδέες που προχωρούν πολύ περισσότερο από την έκθεση της ε, ΕΚΤ. Ε, νομίζω πως οι σωστές στατιστικές θα επιτευχθούν μόνο αν, αν εντείνουμε τις υποπτικές μας αρμοδιότητες. Γι' αυτό και θα πρέπει να γίνονται ευνίδιοι έλεγχοι, ευνίδιε επιθεωρήσεις και όπω ήδη έχει αναφέρει και ο κύριος Κάρας, εγώ θα ήθελα να, επιβεβαιώνονται, να επαληθεύονται οι πληροφορίε που λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα οι στατιστικέ των χωρών τη ευρωζώνη. Όσον αφορά το ψήφισμα, συμφωνώ με το σχέδιο, ιδιαίτερα την έκκληση στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο να ενισχύσουν τι αρμοδιότητε και την απόδοση λογαριασμών, την ευθύνη μάλλον των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, αλλά και την ε, αύξηση των αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ για τον έλεγχο των στατιστικών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμιο όπου η ποιότητα συναντά την ποσότητα. Η ποιότητα, όταν λέμε ποιότητα, μιλάμε για την ποιότητα των στατιστικών. αν δούμε ένα φαινόμενο ας πούμε της ε, πωλήσει κτηρίων ή υποδομών όπου οι κυβερνήσεις πουλούν μια υποδομή και μετά πρέπει να την ξανικιάσουν με πολύ ψηλότερο κόστος ή όταν ε, μιλάμε με συγκεκριμένα τέτοια ταμεία που το έχουμε δει στο παρελθόν ε, όπου αυτά μπαίνουν στο Βέλγιο ας πούμε στον προπολογισμό και μετά βγαίνουν ως υποχρεώσεις. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, αυτό που θα δούμε είναι ότι οι αριθμοί θα είναι πιο αξιόπιστοι, αλλά οι κυβερνήσει θα αρχίσουν να ζουν από το κεφάλαιο που πρέπει, θα πρέπει να το κερδίσουν στο μέλλον. Γενικά συμφωνώ με τον ε, εισηγητή ότι η Eurostat θα πρέπει να γίνει ένα είδος στατιστικού FBI ο εκπρόσωπο της γύρω την εδώ. Ελπίζω να του αρέσουν οι, τα λόγια μου και επειδή είναι και πρώην επικεφαλής ε, του γραφείου μου στην Κομισιόν, είμαι βέβαιος που του αρέσουν τα λόγια μου. Ευχαριστούμε. Hans Peter Martin, μετά από ακούσαμε το FBI. FBA. Ναι, ναι, και εγώ πιστεύω ότι τα στατιστικά δεδομένα αποτελούν ε, και τη βάση, το θεμέλιο κάθε εγχειρήματο και της πολιτικής ζωής και θα πρέπει η πολιτική τάξη αυτό να το ξέρει. Σαφώς και πρέπει να έχουμε αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα και όχι να λέμε διάφορα. Είναι ο κύριος Κάρας ο πιο σκληρά εργαζόμενος και ο πιο απόλυτα δεσμευμένος ευρωβουλευτής από τη χώρα μου. Και σήμερα έχει κάνει εξαιρετική εργασία. Απιστεύω ότι πραγματικά ξεχωρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο συνάδελφός μου. Λοιπόν, αυτά τα οποία μας προτείνει είναι εξαιρετικά, πράγματι εξαιρετικά είναι ένα ε, λίγαν σημαντικό θέμα. Θα ήθελα να συζητήσουμε ε, ενδελεχώς τα θέματα με τη Eurostat, με εκπροσώπους της Eurostat και να δούμε πώς μπορεί η Eurostat να γίνει ακόμα πια πιο ανεξάρτητος φορέας. Βλέπουμε πίσω από τη λέξη Κομισιόν σε παρένθεση να λέει Eurostat που δείχνει ας πούμε μια σχέση εξάρτησης υπάρχουν, έχουν γίνει πάρα πολλά αρνητικά σχόλια για αυτή την ε, ρύθμιση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε έναν ανεξάρτητο φορέα ο οποίος να λειτουργεί ταχύτατα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα, στις πραγματικές ανάγκες. Είμαστε ε, όλοι φιλοευρωπαίοι και αν θυμόσαστε παλιότερα είχαμε μία περίπτωση την περίπτωση αυτή του 2004 όπου οι υπάλληλοι της Eurostat, οι υπάλληλοι της Κομισιόν που ε, συνεχεία έγιναν προϊστάμενοι στο Συμβούλιο ε, άρχισαν τις συζητήσεις των μαζικών λαθών που είχαν υποβληθεί, λαθασμένων στοιχείων μάλλον από την Ελλάδα. Ήταν λοιπόν καταρχάς φιλότιμη υπάλληλοι του Eurostat, εν συνεχεία φιλότιμα στελέχη της Κομισιόν και προϊστάμενοι στο Συμβούλιο που ε, διαπίστωσαν αυτά τα σφαλμένα στοιχεία εάν τα στοιχεία αυτά είχαν γίνει δημόσια, είχαν δημοσιοποιηθεί εξ αρχής, όταν ακόμα βρισκόντουσαν στα χέρια της Eurostat, θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει πολλές πτυχές της ε, καταστροφής αυτής. Πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στους υπαλλήλους, στα στελέχη της Eurostat και να δούμε ε, από τη Eurostat Πού βρισκόμαστε σήμερα με την κρίση του ευρώ. Γι' αυτό δεν συμφωνώ με τον κύριο Σμιτ που λέει ότι τα στατιστικά στοιχεία είναι βαρετά. Εγώ νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να διαμορφώσουμε ένα σενάριο και να είχαμε προβλέψει τι θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει. Δυστυχώς τώρα, τότε, τότε, το 2004, Ποιος ήταν αυτός που εμπόδισε τη Eurostat να εκτελέσει σωστά το ρόλο της. Ήταν όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών. Ήταν οι Υπουργοί Οικονομικών οι οποίοι προέβαλαν όλα αυτά τα προσκόμματα και τελικά επιτρέψαμε αυτή την, ε, το Creative Accounting, ε, την ε, δημιουργική λογιστική και καταλήξαμε σε αυτά τα προβλήματα με την Ελλάδα. Εφόσον λοιπόν διαπιστώνονται λάθη, αυτό που γίνεται δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος είναι υπόλογος. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να μάθουμε από το πάθημα αυτό, πρέπει να συνάγουμε από ε, συμπεράσματα επικοδομητικά για να μπορεί να, να τεθεί ευθύνη και ένα σωστό, μια σωστή ιεραρχία υπόλογου είναι θέματα οργάνωσης, δεν πρόκειται για αστυνομική δύναμη, αλλά πρόκειται για τη σωστή εφαρμογή των αποφάσεών μας, που, είναι πολιτικές. Θέλω λοιπόν ενθαρρύνω του Eurostat να παραμείνει έτσι δραστήρια, να ενεργεί στεναρά, ε, δυναμικά και να μην αποθαρρυνθεί από τα εμπόδια τα οποία σημειώθηκαν στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ε, Έχουμε ακόμα αρκετούς ομιλητές, αλλά είναι ένα σημαντικό θέμα. Η κυρία Τζέρι, Σιλβί Γκουλάρ, η κυρία Σιλκούνη θέλει επίσης να επανέλθει για ένα μικρό. Και εγώ έχω κάτι να προσθέσω. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας αντιμετωπίζει ένα δίλημα εδώ. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Καρά για το ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Όταν πρόκειται για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων ή γενικά για τον οικονομικό, δημοσιονομικό τομέα, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Οι πολίτες περιμένουν από μας ιδέες και πράξεις για να αποφύγουμε πράγματα τα οποία έχουν συμβεί στην Ελλάδα ή στην Ουγγαρία αλλού να μην ξανασυμβούν. Αυτή όμως είναι μια νομοθετική πρόταση και δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε εδώ διατάξεις που δεν έχουν περάσει από ανώτερο επίπεδο. Η ομάδα Φαν μιλάει για την κυριαρχία των κρατών μελών και οι πολιτικές διαπραγματεύσεις έχουν μόλις ξεκινήσει. Δεν μπορεί όμως να κρατήσει για πολύ καιρό αυτή η ιστορία. Ο κόσμος θα γελάει μαζί μας που είμαστε τόσο αργοί. Ούτε μπορούμε και να βιαστούμε για αυτό το θέμα όμως όσο δεν υπάρχει προηγουμένως πολιτική συμφωνία. Όμως, εγώ πιστεύω ότι Ακόμα και με το σημερινό επίπεδο πολιτικής συνένεσης, η έκθεση αυτή δεν φτάνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρκετά φιλόδοξη. Τι έχω κατά νου. Το πρώτο ελληνικό σκάνδαλο το 2004 είχε σαν αποτέλεσμα πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Eurostat να μπορεί να ελέγχει. Απέτυχε αυτή η προσπάθεια. Και τι έχουμε τώρα, μία πρόταση για ερευνητικές εξουσίες. Όμως νομίζω ότι σήμερα είναι πολύ αργά πια. Γιατί πρέπει να διανύσουμε μεγαλύτερη ακόμα απόσταση. Κύριε Λισμίτ, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε για κυρώσεις. Το 2004 είχαμε ήδη λοιπόν τέτοια προβλήματα στην Ελλάδα και τίποτα δεν έγινε ή εν πάση περιπτώσει καμία ουσιαστική αλλαγή δεν έλαβε χώρα στον τρόπο με τον οποίο ε, εξετάζουμε ή επαληθεύουμε τα στατιστικά δεδομένα. Το 2005 στην Ουγγαρία και το 2006 και στην Ελλάδα συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση μέχρι το 2009. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να εισάγουμε ολοκληρωμένες ε, μεταρρυθμίσεις. Το Κοινοβούλιο μπορεί κάλλιστα να ζητήσει από, να ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς το καλό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και πώς είναι δυνατόν να μην ήταν σε θέση να ελέγξουν την κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Όταν πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το Δεκέμβριο, τους ρωτήσαμε κατά πόσο εγνώριζαν τι γινόταν στην Ελλάδα και είπαν ότι ίσως να ξέρανε για το 30%. Ε, δεν φτάνει. Πρέπει να έχουμε εγγύησεις ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη και να κλείσουμε ότι παραθυράκια υπάρχουν. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση, έχει την μεγαλύτερη ευθύνη. Το 2007 η Επιτροπή πρότεινε να σταματήσει η διαδικασία για το υπερβολικό έλλειμμα στην Ελλάδα. Μα αυτό είναι αστείο. Γιατί είχε πάει πολύ μακριά και φτάσαμε σε μια χειρότερη ακόμα κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο αυστηροί από ό,τι είμαστε μέχρι τώρα. Και τα κείμενα πρέπει να είναι πιο αυστηρά και να επιστήσουμε την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ευθύνες της Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Σοφή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στηρίζω ειλικρινά τον εισηγητή. Πιστεύω ότι η προσέγγιση του είναι πολύ σωστή. Εδώ βλέπω ότι διακυδεύεται κάτι πολιτικό πίσω από αυτό το θέμα. Γιατί αν σκεφτούμε μία από τις επικρίσεις που ακούστηκε πιο συχνά και ακούγεται πιο συχνά κατά των Βρυξελών είναι ότι πρόκειται για μια μεγάλη γραφειοκρατία. Ε, λοιπόν, λοιπόν, μια περίπτωση όπου πραγματικά τα κράτη-μέλη, και είναι για να θυμηθώ και αυτό που, λέτε, που είπατε εσείς πριν από λίγο, δεν φταίει μόνο η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη και ακόμα και εκείνα τα κράτη-μέλη που είχαν υποσχεθεί ε, στους πολίτες τους ε, dry comma δηλαδή ότι θα επαληθεύσουν και μετά το κόμμα όλα, δεν το κάνανε. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια περίπτωση εδώ που φέρθηκαν πολύ ελαφρά τα μέλη του Συμβουλίου και έτσι καλλιεργούν έναν λαϊκισμό, έναν, ε, μια στάση κατά των Βρυξελών και κατά της Ευρώπης χωρίς λόγο. Εμείς πρέπει να περάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο όπου η εξέταση των στατιστικών δεδομένων πρέπει να γίνεται σοβαρά και ανεξάρτητα. Μπορεί να μην μιλήσουμε για FBI, αλλά εν πάση περιπτώσει να αλλάξει μέθοδος και το φόβο να τον έχει άλλη πλευρά. Γιατί τα λάθη τα έκαναν οι πρωτεύουσες, δεν τα έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Ο Έντουαρτ. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι, ζητώ συγγνώμη που επανέρχομαι, αλλά ξέχασα να αναφέρω ένα σχετικό θέμα. Τονίζοντας ιδιαίτερα τους ελέγχους και τις εντολές για ελέγχους δεν παραβλέπουμε, παραβλέπουμε ε, σοβαρά την λογιστική μεθοδολογία. Ε, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν διεθνή λογιστικά πρότυπα. Αντίθετα όμως από τον ιδιωτικό τομέα και αυτά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τα σέβονται όλες οι εταιρείες. Αλλά οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν δύο μεθοδολογίες. Υπάρχουν ακόμα χώρες που χρησιμοποιούν ε, αναχρονιστικά συστήματα cash flow και όχι τα σωρευτικά ε, στοιχεία, τα λογιστικά. Ε, οπότε ε, όταν ε, μεταφέρεις τα στοιχεία, τα μεταφράζεις από cash flow σε accrued, κάνεις ε, και τις προσαρμογές όπως τις θέλεις. Δεν το θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε δύο διαφορετικές λογιστικές μεθοδολογίες, θέλουμε ένα ενιαίο σύστημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς αυτό πρέπει να αναφερθεί. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοιες ανισότητες, αν, ανομοιότητες μεταξύ των λογιστικών μεθόδων των κρατών μελών η Πρόεδρος. Και εγώ συγχαίρω τον εισηγητή, έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο και εγώ ως πρόεδρος να πιέσω το Συμβούλιο για το θέμα αυτό και μου φαίνεται ότι είναι απολύτως αναγκαίο να εφαρμόσουμε μία βελτιωμένη και ταχεία μέθοδο ελέγχου και πιστοποίησης. Ε, αυτό πρέπει να είναι προϋπόθεση όποτε θέλουμε να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να υπάρχει ως προϋπόθεση ο σωστός και ταχύς έλεγχος ε, των στοιχείων. Είναι λοιπόν προϋπόθεση για τη σωστή διαχείριση των οικονομικών. Βεβαίω, όταν, όταν λέμε βελτίωση δεν, δεν εννοούμε ότι, ότι αυτό επαρκεί και ότι θα ε, είναι το, το, το, το περισσότερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Ε, πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι ελάχιστη. Είναι ο ελάχιστος παρανομαστής εν ώψη της ελληνικής ε, περίπτωσης. Ε, θα πρέπει οι υποχρεώσεις αυτές να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη-μέλη και να υπάρχει προληπτική δράση, όχι να περιμένουμε κάποιος να ξεπεράσει τα σεμιτά πλαίσια του, του κρατικού ελλείμματος για να παρέμβουμε πρέπει να ξέρουμε στα στατιστικά στοιχεία τι πρέπει να περιλαμβάνονται, δεν περιλαμβάνονται, ε, τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται εκτός ισολογισμού, ποια ακριβώς είναι, σε τι μεγέθη αναφέρονται, γιατί είναι εκτός ισολογισμού. Επίσης πρέπει να ε, να επιτρέψουμε τον έλεγχο των προϋπολογισμών να εφαρμόσουμε μία πολυετή προσέγγιση. Αυτές οι προτάσεις οπωσδήποτε θα αναφερθούν και σε άλλες εκθέσεις. Επειδή ακριβώς έχουμε μία πληθώρα ιδεών σε αυτή την Επιτροπή και θα συναντάμε αυτές τις ιδέες και σε άλλες ε, προτάσεις. Για τις κυρώσεις προτείνουμε στο ψήφισμα να υπάρχει ένα είδος προσωπικής ευθύνης. Σε αυτήν την Επιτροπή μιλήσαμε για προσωπική ευθύνη των διευθυντών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ότι θα υπάρχει το καθεστώς της προσωπικής ευθύνης. όταν αναφερόμαστε στην ανεξαρτησία της Eurostat, από την ε, μία η πρόταση αυτή είναι ελκυστική, από την άλλη πλευρά, όμως, μέσω της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να ασκήσουν περισσότερη εξουσία, έχουν περισσότερη ισχύ. Εγώ προσωπικά δεν έχω καταλήξει στην καλύτερη λύση Ας το σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Πλήρης ανεξαρτησία ή σύμπραξη με την Κομισιόν ή ε, υπό την Κομισιόν. Μέχρι τις 19 του μηνός θα έχουμε και τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας για το θέμα του ψηφίσματος ίσα ίσα μπορούμε να το κάνουμε τον Ιούνιο να το περάσουμε τον Ιούνιο διότι έχουμε συνένεση απόψε, σύμπτωση απόψεων εδώ πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τις δυσκολίες ενός συμβιβαστικού κειμένου, διότι αν καταλήξουμε σε συμβιβαστικό κείμενο θα μπλέξουμε άσχημα. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και να φροντίσουμε να ψηφιστεί τον Ιούνιο. Θα στείλω σχετικά email με αυτήν την παράκλησή μου. Παρακαλώ στο ετών ταχύτερα να διευθετηθούν τα εκκρεμή θέματα για να περάσει, να παρουσιαστεί το ψήφισμα τον Ιούνιο. Υποστηρίζουμε λοιπόν την πρόταση αυτή για τον Ιούνιο και δίνω το λόγο στον εισηγητή εν κατακλείδη. Ευχαριστώ για την εξαιρετική συζήτηση. Μετά από όλες τις ε, συζητήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, ε, βλέπουμε ότι η νομοθετική απόφαση, η νομοθετική πράξη δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες. Υπάρχουν πολλά ακόμα εκκρεμή θέματα. Όμως η πρόταση αυτή και η σημερινή συζήτηση δεν έχουν τη φύση της ερευνητικής επιτροπής. Δεν κάνουμε μία έρευνα προσπαθούμε να, να βελτιώσουμε την πολιτική βούληση με την νομοθετική πτυχή διότι η πολιτική βούληση μεν υπάρχει αλλά δεν έχουμε μπορέσει να τα υλοποιήσουμε όλα αυτά νομοθετικά. Θέλουμε να εκφράσουμε και να εξασφαλίσουμε νομοθετικά τις πολιτικές μας, ε, τα πολιτικά μας πιστεύω και τις πολιτικές μας ε, απαιτήσεις αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολιτικά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε νομοθετικά. Όμως, σας παρακαλώ, κάνω μια έκκληση τουλάχιστον ε, το ψήφισμα αυτό να, περάσει το ταχύτερο για να μπορέσουμε να ενεργήσουμε ευέλικτα δεδομένου ότι αντανακλά την πολιτική μας απόφαση, το πολιτικό μας πιστεύω που σημαίνει ε, ε, ταχύτατη δυνατότητα επέμβασης της Eurostat, αυτόματη ενεργοποίηση των, ε, των αρμοδιοτήτων της Eurostat, ξαφνικές ε, ε, ευνίδιες επισκέψεις ε, στα κράτη-μέλη όπου υπάρχει ανάγκη, απρόσκοπτη συζήτηση με αρμόδιους φορείς και ιδρύματα όπου αυτά κρίνονται κατάλληλα από την Eurostat, και ε, ο, ο έλεγχος, ο σωστός έλεγχος της πιστότητας ε, των στοιχείων που υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά πρέπει να τα τονίσουμε όπως τα εκφράζει το ψήφισμα. Συν η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δίνει γεγονός ότι επί πολλά χρόνια ε, τα πράγματα ήταν στο σκοτάδι, είχαν κουκουλωθεί και αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Και σας παρακαλώ προσέξτε την ε, διαδικασία στην Ολομέλεια μεταξύ προφορικής απόφα... Ε, ερώτησης και ψηφίσματος. Η νομοθετική πράξη εξαρτάται από τη νομική γνωμοδότηση. Αν είμαστε μέσα στη συναπόφαση ή όχι, την περιμένουμε ακόμα όταν θα έχουμε την νομική γνωμοδότηση τότε θα ξέρουμε πώς θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ο, ο εκπρόσωπος της Eurostat θέλει κάτι να προσθέσει σύντομα. Ίσως έπρεπε να σας είχα δώσει το λόγο νωρίτερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω απλώς να τονίσω αυτά τα οποία ήδη είπε ο εισηγητής όσον αφορά τη σημασία αυτής της πρότασης από πλευράς Κομισιόν. Σας είμαστε ευγνώμονες ε, για την ε, προθυμία που δείξατε να εργαστείτε ταχύτατα πάνω σε αυτό το θέμα διότι έχει ιδιαίτερη σημασία και στα συστήματα και στις αγορές. Γι' αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η πρόταση το ταχύτερο δυνατόν. Επίσης θέλω να τονίσω την ε, πολύ καλή συνεργασία που είχα με τις τελευταίες εβδομάδες με μέλη αυτής της Επιτροπής. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις, ε, την πίεση που έχετε ασκήσει και εσείς και τα μέλη της Επιτροπής στο Συμβούλιο. Πράγματι πιστεύω ότι αυτή τη φορά το Συμβούλιο θα είναι πιο ανοιχτό για συνεργασία, θα είναι πιο συνεργάσιμο και πιστεύω ότι θα ολοκληρώσουμε όλες τις διαβουλεύσεις ε, τις ερχόμενες δύο εβδομάδες. Σας ευχαριστούμε και πάλι θαυμάσια συνεργασία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τα μέλη να έχουν υποβάλει μέχρι τη Δευτέρα 7 του μηνός, 4 μετά μεσημβρία τις παρεμβάσεις τους για την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα. Δευτε... για το σχέδιο ψηφίσματος αυτό που θέλουμε να πάει στην Ολομέλεια τον Ιούνιο μέχρι τη Δευτέρα 4 το απόγευμα και μία μέρα παραπάνω για τις ε, τροπολογίες στην νομοθετική πράξη που η προθεσμία είναι 8 Ιουνίου. Συζήτηση τροπολογιών θα γίνει στις 28. Δεν ξέρω αν θα, προλάβουμε τώρα την Ολομέλεια του Ιουλίου. Ευχαριστώ. Θα δώσω το, την Προεδρία στον κύριο Σικλούνα, ο οποίος ε, θα παρουσιάσει την έκθεσή του από, την, ε, τη θέση του Προέδρου. Okay. Okay. We'll see how Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, που είναι η γνωμοδότηση για την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας. Εγώ είμαι ο εισηγητής, ο συντάκτης της γνωμοδότησης, οπότε επιτρέψτε μου να κάνω μερικά σχόλια για αυτό το θέμα. Όπως θα θυμόσαστε, Η αρχική γνωμοδότηση περιλάμβανε προτάσεις ιδιαίτερα που είχαν να κάνουν με τον ορισμό των πράσινων θέσεων απασχόλησης και με τη σημασία που είχε η ταξινόμηση στα στατιστικά δεδομένα αυτών ακριβώς των πράσινων θέσεων εργασίας που δεν εμφανίζονται με τη σημερινή ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων. Έκτοτε πήραμε 10 τροπολογίες, δύο από το ΕΛΚ και τέσσερις από τους πράσινους από τον Φιλίπ Λαμπέρ, δύο από τον Κλούτελ και από την Σοφία Κονή επίσης. θα έρθω στην τροπολογία που αναφέρεται στη γεννητικότητα της ε, αγοράς και που αναφέρεται στις δομικές ελλείψεις. Νομίζω ότι ενισχύει την γνωμοδότησή μας. Το ίδιο έχω να πω και στον κύριο Παντάρ που ενισχύει τον ρόλο της κατάρτισης με το κείμενό του, με την τροπολογία του, όπως επίσης και το ρόλο των επιχειρηματιών. στο τομέα της οικοκαινοτομίας. Οπότε τις θέλω και αυτές τις τροπολογίες. Δύο άλλες τώρα, κλούτε, έχουν να κάνουν με τη σημασία που έχει ο τομέας της απασχόλησης για την υγεία και άλλου είδους κοινωνικές δραστηριότητες. Και υπάρχει κι άλλη μία που αναφέρεται στην ποιότητα των ε, επιχειρήσεων. Έρχομαι τώρα στον Φιλίπ Λαμπέρ. Οι τροπολογίες του έχουν να κάνουν κυρίως με την φορολογία, να μεταφερθεί το βάρος δηλαδή από την εργασία στους πόρους ή μάλλον στις μη ανανεώσιμες πηγές. Μία από αυτές λέει, εκεί που μιλάμε για την ενέργεια, να συμπεριλάβουμε τον όρο μη ανανεώσιμες. Και η άλλη αναφέρεται στον οικολογικό φόρο, carbon tax. Μιλάει για την προετοιμασία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαίσιου προκειμένου να στηρίξουμε την αγορά απασχόλησης. Και προτείνει νέους πόρους μεταξύ άλλων τον οικολογικό φόρο. Εδώ θα μπορούσαμε, Φιλίπ, να συναντηθούμε οι δυο μας και να βρούμε την κατάλληλη διατύπωση. Τώρα θέλω να δώσω το λόγο στους σκιώδες εισηγητές, ώστε να κάνουν οι ίδιοι σχόλια για τις τροπολογίες τους. Ή ό,τι άλλο σχόλιο έχουν να κάνουν. Συνεπώς, πρώτα απ' όλα, ο Φιλίπ Λαμπέρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για τι ανανεώσιμε, ή μάλλον μη ανανεώσιμε. Δεν πρόκειται μόνο για τις πηγές ενέργειας, πρόκειται γενικότερα για τους πόρους. Δεν θα ήθελα να μιλήσουμε μόνο για την ενέργεια. Έχω ένα σχόλιο για την Τανούτα Χιούμπνερ, για τη δικιά της συντροπολογία, δεν νομίζω ότι είναι εδώ. Έχει να κάνει με την κινητικότητα της αγοράς. Καταλαβαίνω τους στόχους της και έχει δίκιο που λέει ότι αν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό πρέπει να δούμε τις δυνάμεις της αγοράς που δεν βρίσκονται πάντα εκεί που τις χρειαζόμαστε. Αλλά η ανησυχία μου εδώ είναι ότι αν είμαστε αρκετά έτσι ευρύς, ασαφείς δηλαδή, προσοχή. Δεν θέλουμε να επαναφέρουμε την αρχή της χώρας προέλευσης. Αν κάποιοι θεωρήσουν ότι για να διευκολυνθεί η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού πριν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο, έχω αντίρρηση. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ υπάρχει αμφισημία. Δεν είναι αρκετά σαφές δηλαδή το κείμενο, γι' αυτό και θα προτιμούσα να απόσχω. Για τις άλλες τροπολογίες και τις δικές μου, αλλά και τις άλλες είμαι σύμφωνος. Πρόεδρος, άλλος που θέλει να πάρει το λόγο για αυτή την γνωμοδότηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχω ένα σύντομο σχόλιο, παρακαλώ, για τις προτάσεις που έχουμε. Ο Φίλιπ ε, Λάμπερτς υπογράμμισε ποιο είναι το πρόβλημα Πράγματι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε ώστε να δώσουμε κίνητρα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να είναι δραστήρες σε μια πιο πράσινη οικονομία και με φορολογικά κίνητρα. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα. Όσον αφορά την κατάρτιση επίσης, εδώ ο κύριος Παντάρ προτείνει κάποιες τροπολογίες που τροποποιούν ριζικά την κατάσταση για να προσαρμοστούμε ακριβώς σε αυτή τη νέα πράσινη οικονομία. Μια άλλη ιδέα είναι η κατάρτιση των ατόμων που ήδη δουλεύουν στις διάφορες επιχειρήσεις. Η πρόκληση είναι μεγάλη. Η αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, στην Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή και πρέπει να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Άρα το προσωπικό των, της αυτοκινητοβιομηχανίας πρέπει να έχει το savoir faire που χρειάζεται, το know-how δηλαδή που χρειάζεται για να μπορέσει να ε, σταθεί στον ανταγωνισμό. Τα αυτοκίνητα, τα κλασικά με τους κλασικούς κινητήρες είναι κάτι διαφορετικό από τα οχήματα που θα έχουμε στους δρόμους μας μετά από λίγο. Και τα στατιστικά δεδομένα εδώ έχουν σημασία. Πρέπει να ξέρουμε ότι στην πράσινη βιομηχανία, ε, ό,τι έχουμε δηλαδή με πράσινη τεχνολογία, να αντικατοπτρίζεται και στα στατιστικά δεδομένα. Οι στατιστικές πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Ναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Σικλούνα. Δεν έχω να συμπληρώσω και πολλά. Τα, οι περισσότερες ε, τροπολογίες είναι καλές, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω κάτι μετά από αυτά που είπε ο Φιλίπ Λαμπέρ όσον αφορά τα φορολογικά κίνητρα. Από την ποια πλευρά μιλάμε για δημόσιους προπολογισμούς που πρέπει να εξηγιανθούν με την εξέβριση νέων πόρων εσόδων και από την άλλη μοιράμε για φορολογικά κίνητρα. Ε, δηλαδή, τι, τι εννοούμε τώρα, περαιτέρω μείωση των φόρων, εδώ θα είχα επιφυλάξεις. Fine. Uh, Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλα σχόλια? Όχι. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλα σχόλια. Οπότε να αναφέρω τις προθεσμίες. Έχουμε ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ στις 22 Ιουνίου και ελπίζουμε ότι μέχρι τότε θα προσπαθήσουμε να τακτοποιήσουμε ε, όλε αυτέ τι αλλαγέ και τι προτάσει, και η ψηφοφορία θα γίνει 14 Ιουλίου στην Επιτροπή την Αρμόδια τη ουσία στην απασχόληση. Ερχόμαστε στο επόμενο θέμα που είναι η εξακρίβωση της νησιότητα των κερμάτων ευρώ και η διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι κατάλληλα για κυκλοφορία. Η συγκεκριτή είναι Μπίνεφ, είναι εδώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Στόχος ε, του προτινόμενου κανονισμού είναι να θεσπίσει διαδικασίες εξακρίβωσης για τα κέρματα ευρώ και για τα, διαχείριση των κερμάτων ευρώ που ε, είναι κατάλληλα για κυκλοφορία. Έτσι θέλουμε να έχουμε κοινέ διαδικασίες για την εξακρίβωση των κερμάτων αλλά και για τους ε, μηχανισμούς ελέγχου της, εξα... διαδικασίας εξακρίβωσης. Κάθε... Ε, Οποιοςδήποτε ασχολείται με αυτή τη διαδικασία επιθυμεί να έχει ένα σαφές κείμενο το οποίο θα θεσπίζει τη διαδικασία εξακρίβωσης των κερμάτων. Από τις τροπολογίες που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι μπορούμε να πούμε πως υπάρχει ένα πνεύμα συνεργασίας η διαδικασία εξακρίβωσης σημαίνει κόστος για τις αρχές και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορούν να έχουν και να, να, χρεώνουν ένα κόστος διαχείρισης ε, Θεωρώ ότι αυτό το κόστος θα πρέπει να αποτελεί επιβάρυνση για τους ιδιώτες και αναφέρομαι στην τροπολογία 41. Στην 43 ε, που έχει υποβάλει ο κύριος Μπάτσο, και που προτείνει ότι μόνο τα κέρματα των 2 ευρώ των, του 1 ευρώ και των 50 λεπτών θα είναι αυτά που θα πρέπει να εξακριβώνονται. Ακατανοώ το κίνητρό του, αλλά δεν δέχομαι αυτό το επιχείρημα για την αλήθεια ότι τα μικρότερα κέρματα των 20 λεπτών ή και τα μικρότερα συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο παραχάραξη, Ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλα τα κέρματα και όλα τα χαρτονομίσματα θα πρέπει να περνούν από διαδικασία εξακρίβωση. Δεδομένης της απουσίας κάποιες απέτησεις εξακρίβωσης για τα κέρματα, οι αρχές δεν θα απαιτείται να αποκαθιστούν τα κέρματα. Καταλαβαίνω πως από ό,τι καταλαβαίνω η διαδικασία είναι διαφορετική. Υπάρχει το θέμα κόστους ωφέλειας η διαδικασία, μάλλον η, τα μηχανήματα εξακρίβωσης κερμάτων δέχονται όλα τα κέρματα. Αυτό σημαίνει πως η εξακρίβωση κερμάτων με μικρή αξία με τα ίδια μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τα υπόλοιπα κέρματα μεγαλύτερης αξίας δεν θα σημάνουν μεγαλύτερο κόστος. Τώρα, όσον αφορά τις άλλες δύο τροπολογίες, 44 και 45 του κυρίου Μπάλτ, που προτείνουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαδικασία εξακρίβωσης. Εγώ πιστεύω πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην εξακρίβωση μέσω μηχανήματος ή την ε, διαχειρός. Η 46 της κυρίας Οκονή ε, λέει ότι θα πρέπει να προβλέπεται μια λογική προθεσμία ε, εντός, για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1. Εγώ υποστηρίζω αυτή την τροπολογία και ελπίζω πως θα φτάσουμε σε συνένεση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Σε σχέση με την ε, ακύρωση της χρήσης κάποια μηχανής εξακρίβωσης λόγω βλάβης Δεν νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ισχύσει και αναφέρομαι στην ε, τροπολογία 47. Υποστηρίζω αντίθετα την 48 ε, και σε σχέση με το δικαίωμα του κράτους μέλους να, ζητήσει εγγυήσεις από εκείνα τα θεσμικά όργανα που εξακριβώνουν τα κέρματα και την απέτηση για σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό. Τώρα, για την κατάρτιση του προσωπικού, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνολογίας και Επιστημών η αρμόδια αρχή για τις ε, τροπολογίες 49 και 45 κατά τη διάρκεια ε, διαβουλεύσεων με ειδικούς της Όλαφ κατάλαβα ότι υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου ε, κλέβουν τα φορτηγά μεταφοράς κερμάτων και εκεί εκλείονται αέρια ή οσμές. Ε, αυτά οφείλονται στην, εξαιρετική, στην υπερβολική χρήση των ουσιών που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των κερμάτων και γι' αυτό όταν υπάρχει λόγος να πιστεύει κανείς ότι υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, τότε τα ε, τέλη χειρισμού, διαχείρισης θα πρέπει να συμπληρώνονται από ένα επιπλέον 20% της αρχικής αξίας. Για την παράγραφο 9 ε, θέλω να, να προτείνω το εξής ε, κείμενο. Να τα κέρματα θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί και να στέλνονται στις αρμόδιες αρχές. Και αυτό για προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια. Από τεχνική άποψη, όλα τα μηχανήματα εξακρίβωσης ε, απορρίπτουν τα κέρματα που είναι κατάλληλα για κυκλοφορία και τα κέρματα που πιστεύετε ότι είναι παραχαραγμένα. Πλαστά. Αυτά συσκευάζονται και στέλνονται στην αρμόδια εθνική αρχή που τα αναλύει και αποφασίζει ποια μηχανήματα, ποια κέρματα είναι πλαστά και ποια όχι. Από λειτουργική άποψη, βιομηχανία χρειάζεται την εξή ε, αποσαφήνιση. Τα σωστά κέρματα και αυτά τα οποία έχουν, είναι πλαστά θα πρέπει να συσκευάζονται από κοινού όταν στέλνονται στην αρμόδια αρχή και δεν πρέπει να ξεχωρίζονται σε διαφορετικές συσκευασίε. Τροπολογία 51. Θεσπίζει μια προθεσμία για την 31η Δεκεμβρίου του 2015 Μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει πρόταση. Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω τα, τα, τα, τους ευρωβουλευτές ε, που είναι εδώ παρόντες ότι αυτό είναι ένα θέμα που έχει επανειλημμένως ε, ε, συζητηθεί. Δεν υπάρχει συνένεση ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες και τα κράτη για το θέμα αυτό. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι ακόμα και αν υπάρξει συνένεση σε τεχνικό επίπεδο για τεχνικούς ορισμούς, για τα μηχανήματα δηλαδή που είναι σε θέση να αξιολογήσουν όλες τις παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά των κερμάτων, το κόστος θα ήταν υπερβολικά ψηλό. Τα αφήνω σε εσά να αξιολογήσετε τις τροπολογίες και προσβλέπω στην δική σας κατανόηση και συνεργασία. Θα ζητήσω τώρα, θα ρωτήσω τώρα τους ε, σκέδου ηγητέ να μας πούν τι απόψει του. Έχουμε πρώτη Σοφία Κονή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα πρέπει να συγχαρώ τον εισηγητή για την ποιότητα της δουλειάς του και για τον τρόπο με τον οποίο ε, μας ε, μάλλον ηγήθηκε τη συζήτηση, καθώς και για την δυνατότητα, την, τα καταπληκτικά του γαλλικά. Ε, να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου που ήταν ιδιαίτερα ανοιχτή και έδειξε μεγάλη διαθεσιμότητα. Εγώ έχω καταθέσει τρεις τροπολογίες, την 41, που λέει ότι κάθε θεσμικό όργανο που κάνει εξακρίβωση κερμάτων σε ευρώ μπορεί να ζητήσει ε, τέλη σε σχέση με τη διαδικασία εξακρίβωσης, ωστόσο αυτά τα έξοδα θα πρέπει να βαραίνουν ιδιώτες. Φυσικά εδώ πρόκειται για μια τροπολογία που εξασφαλίζει πως οι δαπάνες, τα έξοδα της εξακρίβωσης δεν θα βαραίνουν ιδιώτες. Ε, η 46 που λέει ότι η Κομισιόν δημοσιεύει τις κατευθύνσεις γραμμές σε, μια λογική, σε ένα λογικό χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύω αυτού του κανονισμού ώστε να εγγυηθούμε την τεχνική εφαρμοσιμότητα των διατάξεων της παραγράφου 1, ώστε να ζητήσουμε δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν να δημοσιεύσει τις σχετικές της παρατηρήσεις. Και έπειτα, Εάν υπάρχουν κέρματα που έχουν ευλαθεί από επικίνδυνα προϊόντα σε τέτοιο βαθμό που να θεωρείται ότι, ότι αυτά αποτελούν κίνδυνο για τους ανθρώπους που τα χειρίζονται, εκεί θα πρέπει να επιβαρυνθούν με περαιτέρω τέλη ε, που αντιστοιχεί στο 20% της ονομαστικής αξίας των εν λόγω κερμάτων. Εδώ ίσως μιλάμε καλύτερα για κατεστραμμένα κέρματα τα οποία μπορεί να βλάψουν την εικόνα του ευρώ. Αυτά για την 49. Τώρα, για την 43 που στοχεύει στο να αποκλείσει από την εξακρίβωση τα κέρματα με χαμηλότερη αξία, κάτω δηλαδή από τα 50 λεπτά, καταρχήν αντίθετη με τον κανονισμό του 2001, μια τέτοια πρόταση, και έπειτα βάζουμε στην άκρη τα κέρματα των 20 λεπτών και των 10 λεπτών και δίνουμε κακό μήνυμα προς τους παραχαράκτες αφήνοντάς τους να φαντάζονται ότι θα τους αφήσουμε να δουλεύουν πάνω σε αυτά τα κέρματα. Ίσως θα πρέπει αυτά να τα συζητήσουμε με τον συνάδελφο που συνέταξε αρχικά αυτήν την τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έλαβε υπόψη της τροπολογίες μου για την διαχείριση, για το πώς θα διαχειριστούμε τα κατάλληλα νομίσματα και επίσης για την υιοθέτηση κοινών εκπαιδευτικών προτύπων η τροπολογία μου για τα μηχανήματα τα οποία έχουν χαλάσει, τι θα κάνουμε με αυτά. Ε, καταλαβαίνω ότι είναι σημαντική η τροπολογία αυτή. Εν μέρη καλύπτεται από το αιτιολογικό, από τα εκτιμώντα πέντε και είναι το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Τεχνολογικό Κέντρο που είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιληφθεί αυτή η, αυτή η πρόταση στην έκθεση. Η ιδέα είναι πώς θα μεταχειριστούμε τις ε, ε, χαλασμένες μηχανές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κατάλληλη διαδικασία. Τι θα γίνει αν αυτά τα μηχανήματα χαλάσουν και δεν τα χρειαζόμαστε πια. Πρέπει να προλάβουμε μια κατάσταση όπου τα μηχανήματα αυτά μπορεί να πέσουν σε λάθος χέρια και να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση ε, παραχαραγμένων ε, νομισμάτων. Ευχαριστώ. Επειδή προέρχομαι από μια χώρα εκτός Ευρωζώνης, ε, καταλαβαίνω ότι όταν μιλάω πρέπει να είμαι εξαιρετικά ευαίσθητη στα θέματα αυτά. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την έκθεση. Είναι σαφές ότι ο εισηγητής έχει δουλέψει επιμελώς. Έχει εξετάσει όλες τις πτυχές του προβλήματος και εμά μας ανησυχεί βεβαίως η τροπολογία που λέει ότι δεν θα χρειάζεται εξακρίβωση σε ένα κέρμα αξίες λιγότερο των 50 λεπτών. Ε, αυτό μπορεί να δώσει κίνητρα στην περαιτέρω παραχάριξη των μικροτέρων κερμάτων. Αυτή είναι μόνη μας επιφύλαξη, διαφορετικά συμφωνούμε με αυτά που είπε ο εισηγητής και άλλοι. Λίγες επιφυλάξεις έχω και για την τροπολογία 21. Αυτό ίσως οφείλεται στην, ίσως οφείλεται στην αγγλική μετάφραση όπου αναφέρεται το θέμα ενός φορέα ο οποίος ήταν υπεύθυνο για την εξακρίβωση αλλά δεν σεβάστηκε τους κανονισμούς και ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διόρθωση των εσφαλμένων διαδικασιών που εφάρμοσε αυτός ο φορέας μέσα σε μια ευλογή χρονική περίοδο. Δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί σωστά στα αγγλικά, αλλά θα την ξανακοιτάξω αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ. Ε, η Κομισιόν έχει ο κύριος Ξε, Ξενάρης κάτι να πει. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να, ε, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ντίνεφ για όλη αυτή τη δουλειά που έκανε και όλες τις πρακτικές και μηχανολογικές λεπτομέρειες τις οποίες εξέτασε. Ε, πραγματικά πρέπει να σας συγχαρώ για αυτή την ε, προσπάθεια. Η γενική κατεύθυνση της ε, γνωμοδότησης και των τροποποιήσεων όπως αξιολογήθηκαν από τον κύριο Μπίνεφ συνάδουν με τη γενική μας προσέγγιση. Ευχαριστώ επίσης και και όλους τους συζητητές και τα άλλα μέλη του Κοινοβουλίου που υπέβαλαν τροπολογίες. Επίσης και εγώ έχω επιφυλάξεις για, για την πρόταση να περιορίσουμε την ανάγκη εξακρίβωσης στα κέρματα υψηλότερης ονομαστικής αξίας ε, πάνω από τα 50 cents. Πιστεύω ότι αυτή η πρόταση δεν ε, συμβαδίζει με το μήνυμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε κατά ε, των παραχαρακτών. Έχω δύο πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις. Καταρχάς τα χαλασμένα μηχανήματα. Αυτό βασίζεται, αυτό αναφέρεται σε μία τροπολογία του κυρίου Παντά ε, πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι κάνουμε με τα χαλασμένα μηχανήματα. Εάν το μηχάνημα αυτό δεν μπορεί πλέον να εκτελεί την ε, εργασία εξακρίβωσης, ίσως να πουληθεί σε κάποιον που δεν κάνει εξακρίβωση, εργασίες εξακρίβωσης. Παραδείγματος χάρη σε ένα περίπτερο ή σε ένα εκκλησιαστικό φορέα ή σε κάποιο άλλο ίδρυμα που δεν υποχρεώνεται να κάνει τη διαδικασία εξακρίβωσης. Άρα λοιπόν αντί να καταστρέψουμε αυτά τα μηχανήματα και παρόλο που δεν είναι σε θέση πλέον να εκτελούν τον αρχικό σκοπό τους, ίσως μπορέσουμε να τα πουλήσουμε σε ιδιώτες, σε άλλους φορείς, που να τα λειτουργήσουν διαφορετικά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να καταστραφούν αυτά τα μηχανήματα. Το η δεύτερη μου παρατήρηση αναφέρεται στην πρόσθετη παρατήρηση που έκανε ο κύριος Μπίνεφ όσον αφορά τη συσκευασία, το πακετάρισμα των ακατάλληλων νομισμάτων μαζί με παραχαραγμένα κέρματα. Και πάλι ε, το εκτιμώ ιδιαίτερα και το θαυμάζω για το πώς κατανόησε αυτά τα θέματα. Είναι σημαντικό αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε ακόμα λύση. Ο κύριος Μπίνεφ ε, ε, λέει ουσιαστικά ότι αντί η εταιρείε να διαχωρίζουν όσο καλύτερα μπορούν τα κατάλληλα από τα παραχαραγμένα, ας τα συσκευάσουν όλα μαζί και να τα στείλουν στον αρμόδιο φορέα, ώστε ο αρμόδιος φορέας να κάνει αυτή τη ε, δουλειά. Δύσκολη αυτή η συζήτηση, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να απαντήσουμε σήμερα Έχω τις δικές μου ιδέες, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε μια κατάλληλη διατύπωση, η οποία να καλύπτει τις επιφυλάξεις και ταυτόχρονα δεν θα επιβαρύνει με πρόσθετες υποχρεώσεις τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι εν τέλει θα βρεθούν υποχρεωμένοι να ξεχωρίζουν ένα-ένα τα κατάλληλα νομίσματα για να βρουν εκατοντάδες ακαταλλήλων νομισμάτων για να βρουν 5-10 παραχαραγμένα. Ε, ξέρω ότι το πρόβλημα αυτό είναι πραγματικό και πρέπει να βρούμε μία λύση. Γενικά όμως επαναλαμβάνω ότι ευχαριστώ τα επικοδομητικά σχόλια τα οποία ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ξενάρη, ευχαριστώ και τον εισηγητή λέει ο πρόεδρος, στην Οίκον, στην Επιτροπή μας 22 Ιουνίου θα γίνει ψηφοφορία για την Ολομέλεια ε, του Σεπτεμβρίου. Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Υποθέτω ότι δεν θα έχετε τίποτα άλλο να σχολιάσετε. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση το τελευταίο θέμα στην μερίσια διάταξη είναι οι πολιτικέ απασχόλησης των κρατών μελών. Κατευθυντήριε γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησει των κρατών μελών. Δεύτερο μέρος των ενσωματωμένων ο, ε, κατευθυντηρίων γραμμών του 2020. Και δίνω το λόγο στον κύριο Μάρτιν που είναι συγγητή. Ευχαριστώ. Είμαστε στο τέλος της ε, συνεδρίασης, τελικά θα μείνουμε δυο μας. Έχω ε, κατανόηση ότι η Επιτροπή αυτή έχει πολλές άλλες προτεραιότητες, γι' αυτό θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Εδώ πρόκειται για την απόφαση του Συμβουλίου δεύτερο τμήμα των κατευθυντηρίων γραμμών για την Ευρώπη 2020. Ε, δεν εξεπλάγει όταν τέλο πάντων είσαι αυτό το θέμα σε τέτοια διάσταση. καταρχά πρέπει βεβαίως να πούμε ότι η Λισαβόνα δεν λειτουργήσε, αυτό το λαμβάνω υπόψη από την αρχή. Δεύτερον πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένε διαδικασίες, ειδικά η Λισαβόνα μας έδειξε ότι αλλάζουμε συνεχώ τι παραμέτρου, στο τέλο δεν καταλήγουμε πουθενά. Το αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Γι' αυτό η τροπολογία μου 7 εκφράζει ακριβώς αυτά τα, αυτά τα αρνητικά συμπεράσματα. Επίσης έχω τη φιλοδοξία και πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε το θάρρος να αυξήσουμε τους στόχους μας, να τους ανεβάσουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο για να μπορέσουμε να μειώσουμε την ανεργία και τον αριθμό των ανέργων μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης 2020 και επίσης να σας ε, θυμίσω ότι δεν χρειαζόμαστε μόνο συγκρισιμότητα στα στατιστικά αλλά και στα χαμηλότερα επίπεδα, ειδικά στην εκπαίδευση, ειδικά ε, στην εκπαίδευση δασκάλων, καθηγητών. Ε, εκεί υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά τη διακίνηση ε, καθηγητικού προσωπικού, ε, προσφορά υπηρεσιών στον ε, τομέα της παιδείας. Αυτά τα καλύπτονται στην τροπολογία 11 και είμαι και της άποψης ότι θα πρέπει ιδιαίτερα ταλαντούχοι να τύχουν ιδιαίτερης μεταχείρισης, να τους βοηθήσουμε η τροπολογία 14 αναφέρεται στις δαπάνες παιδείας και ζητάει να καλύπτουν τουλάχιστον 6% του ΣΑΕΠ. 6% του ΑΕΠ. Αυτό το 6% ε, δεν μου ήρθε με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, αλλά βασίζεται στην έκθεση του ΟΣΑ και ε, αυτά, αυτό το 6% το έχει ξεπεράσει προς το παρόν η Δανία με 7,2%, η Σουηδία επίσης είναι πάνω από το 6%, το Βέλγιο επίσης, αλλά η Γερμανία περιέργως ούτε 5% του ΑΕΠ δεν είναι δαπάνες για την παιδεία. Ε, το 6% λοιπόν είναι ο μέσος όρος όλων των κρατών του ΩΣΑ και αν κοιτάξουμε τους στόχους της Λισαβόνας είναι πραγματικά εντυπωσιακό, εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία έχουν πολύ μεγαλύτερες ε, δαπάνες ε, αναλογικά με το ΑΕΠ άρα λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς αυτή την κατεύθυνση και τέλος πιστεύουμε ότι πέραν της ανεργίας των νέων πρέπει να έχουμε τη φιλοδοξία και στον ορισμό της φτώχειας να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να αυξήσουμε ε, ε, και να, και να μειώσουμε το ποσοστό της στόχης κατά 25%. Είναι, είναι ντροπή που αυτή τη στιγμή ακόμα 80 εκατομμύρια ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Πρέπει να το μειώσουμε το ποσοστό αυτό κατά 25% τουλάχιστον. Αυτά είναι τα βασικά που είχα να πω για τις τροπολογίες. Ευχαριστούμε. Έχει... Θέλει κανείς το λόγο. Υπερβάνς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μπορώ να σχολιάσω τη γνωμοδότηση της Πέτερ Μάρτιν τέτοια ώρα. Σχεδόν κανείς δεν είναι στην αίθουσα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ανησυχώ και που θλίβομαι γιατί εγκαταλείπει η Επιτροπή μας όλα τα μακροοικονομικά θέματα. Προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να παρέμβει μακροοικονομικά, δεν έχουμε τίποτα σχεδόν πια στη διάθεσή μας. Εντάξει, δεν πρόκειται να σας βγάλω λόγο τώρα μπροστά σε τρεις ανθρώπους, αλλά μια που μου δίνετε ευκαιρία θα σας το πω. Μια παρέμβαση είναι, δεν, είναι, δεν βγάζω λόγο. Η απόφαση που πήρε η Επιτροπή μας είναι πάρα πολύ σοβαρή. Η κρίση στην Ευρωζώνη σήμερα δεν είναι η κρίση του ελληνικού χρέους. Η κρίση της Ευρωζώνης σήμερα είναι πεποίθηση των αγορών ότι δεν υπάρχει πιλότο αεροπλάνο. Ότι η σταθερότητα δεν αποτελεί επαρκές οικονομικό και αποτελεσματικό μέσο. Η σταθερότητα τιμών. Χρειαζόμαστε λοιπόν οριμότητα στον τομέα της οικονομικής πολιτικής ότι λοιπόν μπορεί να μοιάζει με εξάντε συντονισμό, είναι αναγκαίο. Το μόνο μέσο όμως που έχουμε σήμερα μπροστά μας που είναι αναποτελεσματικό, απογοητευτικό, ακαδημοκής, θεωρητικό δηλαδή. Όμως είναι το μόνο μέσο εξάντε που έχουμε και είναι οι μεγάλες κατευθυντήριες γραμμές. Και η Επιτροπή μας τι αποφασίζει να μην ασχοληθεί με τους προσανατολισμούς αυτούς, με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Μα αυτή η απόφαση για μένα είναι απίστευτη. Ξέρω, υπήρχε περιορισμός χρόνου, ήταν 27 Απριλίου, το Συμβούλιο έτσι κι αλλιώς θα είχε αποφανθεί χωρίς να μας ακούσει. Αυτός όμως δεν είναι λόγος για να παραιτηθούμε. Για μένα η απόφαση αυτή, και είναι δύσκολο να το πω. Ήμουνα πριν πρόεδρος και δεν είναι ότι θέλω να είμαι επικριτική απέναντι στην καινούρια προεδρία της Επιτροπής αυτής. Δεν το λέω γι' αυτό. Έχουμε τόσο σοβαρά θέματα και εμείς κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μα δηλαδή δεν πρέπει το Κοινοβούλιο να παρεβαίνει σε αυτά. Κάνουμε ένα ψήφισμα για την οικονομική διακυβέρνηση στην Ολομέλεια. Ναι, μπλα μπλα μπλα. Με ειλικρινά Εντάξει, καταλαβαίνω ότι φαίνεται, ακούγεται σουρεαλιστική τέτοια ώρα, τέτοια λόγια η δικιά μου παρέμβαση εδώ, αλλά ναι, το ξέρω ότι έχουμε μια γνωμοδότηση για τις κατευθυντήριες γραμμές. Ε, εντάξει, θα μας ακούσει η Επιτροπή Απασχόλησης. Αν όμως εμείς έχουμε να πούμε κάτι γι' αυτό, δεν έχουμε να πούμε για τους μεγάλους οικονομικούς προσανατολισμούς. Ε, φέραμε τα πάνω κάτω. Τι είναι αυτά. Ουρλιάζω θα προτιμούσα να είχαμε περισσότερου εδώ να μ' ακούσουν, αλλά ελπίζω ο Προεδρεύων εδώ να περάσει το μήνυμά μου. Thank you Ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα λόγια. Ναι, νομίζω ότι πολλοί σας στηρίζουν. Λοιπόν, ε, θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Κρίξεν. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχήν, ευχαριστώ το Χάνς Πίτερ Μάρτιν η πρόταση αυτή γνωμοδότησης είναι επικοδομητική. Μπορεί να μην συμμερίζομαι όλες του τις ε, απόψεις, παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι ένα καλό σημείο ε, κίνησης για συζήτηση. Μιλάει ο συγητής για τους σφαιρικούς στόχους υπέρ της απασχόλησης, καταπολέμηση της ανεργίας. 80% δεν ξέρω αν είναι εφικτός στόχος, και δεν είμαι και σίγουρος ότι είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για μείωση 30% στη φτώχεια. Αλλά βέβαια τέτοιους στόχους πρέπει να συζητήσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι φυσιολογικό να βάζουμε ψηλούς στόχους, αλλά και στόχους που να αντικατοπτρίζουν αυτό που μπορούμε να πετύχουμε, αυτό που είναι εφικτό. Το να δουλεύουμε με μη ρεαλιστικούς στόχους δεν ε, βοηθάει πολύ, μπορούμε όμως να τους συζητήσουμε. Θέλω να αναφέρω πέντε σημεία. Πρώτον, χρειάζεται καλή ισορροπία για τη στρατηγική εξόδο από την κρίση. Χρειαζόμαστε παγίωση των δημοσιονομικών ε, των κρατών μελών. Από την άλλη μεριά θα ήταν αρνητικό να δούμε να διαλύονται τα μέτρα αυτά έξοδο από την κρίση πολύ γρήγορα. Γιατί έτσι θα σταματήσει η ανάκαμψη. Δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο λοιπόν, να μην σταματήσουμε την ανάκαμψη. Δεύτερον, πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την απασχόληση. Είναι μακροχρόνιος βέβαια στόχος. Όλοι, άντρες και γυναίκες, πρέπει να απασχολούνται στο ίδιο επίπεδο. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζονται ανανομένες προσπάθειες που να διασφαλίζουν στις γυναίκες τι ίδιες ευκαιρίε στην αγορά εργασίας, όπως γίνεται και με τους άντρες. Τρίτον, κεντρική σημασία θέμα είναι οι διορθωτικές μεταρρυθμίσει στα κράτη-μέλη να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε η ανάπτυξη να οδηγήσει σε μεγαλύτερη απασχόληση. Η ανάπτυξη δηλαδή να είναι τέτοια που να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόληση στην πραγματική οικονομία. Εάν η δημιουργία θέσεων απασχόλησης δεν είναι κεντρικό θέμα στην ανάπτυξη, θα καταλήξουμε με υπερβολικά μεγάλη ανεργία, χωρίς να μπορούμε να τη μειώσουμε με τίποτα. τον. πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο κλειδί των ε, κοινωνικών εταίρων στην αγορά εργασίας και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών επίσης. Η πολιτική απασχόληση των κρατών μελών θα πετύχει μόνο εφόσον ξεκινήσουμε από τη σύλληψη της πολιτικής αυτής και συμπεριλάβουμε εκεί την, ε, τις νέες θέσεις απασχόλησης και σεβαστούμε τους κοινωνικούς εταίρους και έχουμε συλλογικές συμβάσεις ώστε να διαπραγματευτούμε για τις συνθήκες εργασίας. Πρέπει μαζί να γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό και για ολόκληρη την κοινωνία. Πέμπτον, στις συζητήσει για τα δημοσιονομικά των κρατών μελών δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επενδύσεις είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την απασχόληση και για τη συνοχή. Και αυτό πρέπει να φαίνεται στον προπολογισμό. Λιγότερη ανεργία, λιγότερη φτώχεια σημαίνει λιγότερες κοινωνικές δαπάνες. Άρα περισσότερα έσοδα για τις χώρες. Αυτό είναι ένας κανόνες που πρέπει να τον ε, δεχτούμε όλοι. Υπάρχει λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας. Εξετάζουμε αργά την έκθεση αυτή. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε την πρόταση του κύριου Μάρτιν γιατί αποτελεί ένα πολύ καλό σημείο κίνησης για συζήτηση. Ευχαριστώ. Έφερε. Ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ. πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα συγχαίρω που καταφέρνετε να τελειώσετε τη συνεδρίαση στην ώρα τη και λυπάμαι που δεν ήμουν εδώ εξ αρχή. Συγχαίρω και τον εισηγητή για την γνωμοδότηση αυτή. Για να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξασφαλίσουμε μια δυναμική επιχειρησιακή ατμόσφαιρα, ένα περιβάλλον που να ενισχύει τον ε, θεμητό και ελεύθερο εμπόριο, το θεμητό ανταγωνισμό, ένα υγιές περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί όπως ξέρουμε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν και τις πιο πολλές θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να ορθολογήσουμε όλο το πλαίσιο λειτουργίας τους και να η εργατική μας να είναι ευέλικτη. Όλη αυτή η ακαμψία της εργατικής νομοθεσίας έχει δημιουργήσει ένα δυσμενές περιβάλλον για την αγορά εργασίας και θα πρέπει να μειώσουμε και την, ε, ε, το παρεμβατικό πλαίσιο του δημοσίου, των κυβερνήσεων και των κρατών βλέπουμε ότι το κόστος της εργασίας με το τεράστιο ρυθμιστικό πλαίσιο που έχουμε συνεχώς αυξάνεται και έτσι λιγότεροι άνθρωποι απασχολούνται για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ε, έναντι του, του άλλου του υπόλοιπου κόσμου πρέπει να αυξήσουμε την προσπάθειές μας για καινοτομίες πρέπει να βελτιώσουμε την παιδεία χρειάζεται η σύναψη νέων συμφωνιών συνεργασίας ε, μεταξύ ε, των οικονομικών τομέων και των πανεπιστημίων και χρειάζονται και περισσότερες επενδύσεις. Πρέπει επίσης να διαχειριστούμε τις δημογραφικές αλλαγές. Πρέπει οι άνθρωποι να εργάζονται περισσότερο. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα ε, μια υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης to help Και συμφωνούμε με τον κύριο Μάρτιν ότι μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των εργαζομένων και ταυτόχρονα να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Αυτά θα επιτύχουμε με τη μείωση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Δεν θέλουμε νέο, πολλούς καινούριου στόχους, ιδιαίτερα όταν οι στόχοι αυτοί δεν έχουν αξιολογηθεί όσον αφορά τις επιπτώσεις τους. Δεν υπάρχει λόγος να παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα, να είμαστε διάσπαρτοι δηλαδή από εδώ και από εκεί, χωρίς να έχουμε την δυνατότητα εποπτείας και αξιολόγησης Πιστεύω ότι αυτή η γνωμοδότηση θα βοηθήσει ιδιαίτερα την Επιτροπή Επασχόλησης. Σας ευχαριστώ κύριε Φόξ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, ζητώ από τον κύριο Μάρτιν να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ θερμά. Συμφωνώ με όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν. Συμφωνώ μαζί σας ε, κύριε εισηγητά. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει ένα σαφέστατο μήνυμα για τις μακροοικονομικές του προθέσεις και, προσδοκίες. Δεν λέω ότι εδώ ανακαλύπτουμε την ε, πυρίτιδα, αλλά ε, πρόκειται για τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που θέλουμε να υλοποιηθούν. Ευχαριστώ και τους, ε, τα μέλη τα οποία έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Πολλές φορές βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι. Ε, πήγαν στο φεγγάρι, γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Και εγώ προτιμώ λιγότερους στόχους, αλλά δυστυχώς ε, μας επιβλήθηκαν, μας επιβλήθηκαν από το Συμβούλιο. Εγώ προσπαθώ να περάσει τουλάχιστον το 6% στην παιδεία. Δεν πιστεύω ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξος αυτός το στόχος, ο στόχος. Και ο κύριος Φόξ μπορεί να το ελέγξει αυτό, μπορεί να, το, να, δει αυτό το στοιχείο στην έκθεση του ΩΣΑ. Το 6% σας είπα, το λέει συγκεκριμένα ΩΣΑ, έχω μάλιστα και το απόκομα εδώ, Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα μέλη. Σας εύχομαι ε, καλή, καλό Σαββατοκύριακο, ιδίω αυτούς που ήδη έχουν φύγει, οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί. Ο Πρόεδρος, προθεσμίες, ημερομηνίες, 8 Ιουνίου, ε, προθεσμία τροπο, υποβολής τροπολογιών, συζήτηση των τροπολογιών 21 Ιουνίου, ψηφοφορία στην οίκον 22 και Ολομέλεια 1η Σεπτεμβρίου. Ο, τελική ψηφοφορία 14 Ιουλίου, ολομέλεια, 1η ε, Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Στα διάφορα, επόμενη συνεδρίαση στο Στρασβούργο, Δευτέρα 14 στι 7 το απόγευμα και μετά Βρυξέλλες την Δευτέρα, 21η το απόγευμα και Τρίτη όλη τη μέρα, 22 Ιουνίου. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.